Συνάδελφοι καθίστε. Σας καλωσορίζω όλους. Θα ξεκινήσουμε χωρίς καθυστέρηση. Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης μπορεί να θεωρηθεί δεκτό εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Τα πρακτικά της 11ης και 25ης Ιανουαρίου είναι ήδη στα έγγραφά σας, στο φακελό σας. Αν δεν έχετε παρατηρήσει, θεωρούνται δεκτά. Περνάμε στο σημείο 3. Υπάρχει διερμηνία για όλες σχεδόν τις γλώσσες. Σα Ουγγρέζε, Λιτουάνο, Πολάκο, Βούλγαρο και Ρουμένο. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει αναμετάδοση στο διαδίκτυο της συνεδρίασης τα αποτελέσματα της συνεδρίασης των, συντονιστών στις 26 Ιανουαρίου έχουν αποσταλεί σε όλα τα μέλη και υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά όρια για να εκφράσετε τα σχόλιά σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Γραμματικάκη μπόρεσα να πάρω μέρος σε μια μεγάλη συνάντηση ε, θα έλεγα στην Θεσσαλονίκη ε, για τα σε εισαγωγικά για την ημέρα όπου ε, εορτάστηκε ο Αριστοτέλης θα ήθελα επίσης να σας μεταφέρω ένα, αυτά τα σχετικά με τον, με έναν Ιταλό ερευνητή από το Πορντενόνε, νέο στην ηλικία, ο οποίος πήρε το βραβείο των νέων ερευνητών για το 2014 και δυστυχώς με μια ομάδα ερευνητών είχε πάει στην Αίγυπτο και ε, δολοφονήθηκε, βασανίστηκε, κανένας ακόμα δεν ξέρει το γιατί και θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο το συγκεκριμένο νέο ερευνητή γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ε, μαχητής για μια ακέραιη μορφή έρευνας, για μια δημοκρατική μορφή έρευνας και δεν θα πρέπει να τον ξεχάσουμε. Και να εκφράσουμε επίσης τα συλληπιτήριά μας και προς την οικογένειά του που έχασε ένα τόσο σημαντικό νέο άνθρωπο, είναι μια οικογένεια σχετικά φτωχή, αλλά ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει εξαιρετικές σπουδές και στο Κέμπριτς και όχι μόνο στην Ιταλία. Χθες στη Ρώμη έγινε κάτι αρκετά σημαντικό. Υπεγράφει μια συμφωνία της Ιταλικής κυβέρνησής μου Θυμάστε ότι είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό ε, κάποιες ε, συζητήσεις για την αποτροπή της καταστροφής της διεθνούς κληρονομιάς στα πλαίσια της UNESCO. Και στο Συμβούλιο ε, της UNESCO τον Οκτώβριο ξεκίνησε η προσπάθεια για τους κιανόκρανους του πολιτισμού ε, θα υπάρξουν διευκρινήσεις γύρω από τη συμφωνία αυτή. 60 ε, μέλη θα έχει η δύναμη αυτή σε μία πρώτη φάση, 30 θα είναι αστυνομικοί και οι υπόλοιποι εμπειρογνώμονες θα υπάρξει μια έδρα αυτής της ε, ομάδας των πολιτιστικών κιανοκράνων ε, στο ε, Τωρίνο και η Μπόκοβα θύμισε επίσης ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πρώτο το οποίο έχει ζητήσει τη δημιουργία αυτού του σώματος και υπάρχει πρόταση και άλλες χώρες να υπογράψουν μια τέτοια συμφωνία διμερή με την UNESCO και ίσως και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να παρουσιάσει μια τέτοια έκκληση στον ΟΗΕ. Είναι η κατάληξη μιας θεσμικής πρωτοβουλίας, μιας πολιτικής πρωτοβουλίας. Τον Απρίλιο θυμίζω ήμασταν το πρώτο κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ζήτησε να υπάρξει αυτό το σώμα των πολιτιστικών ε, και ανοκράνων. Λοιπόν και τώρα φτάνουμε στις ψηφοφορίες. Η πρώτη ψηφοφορία είναι η έκθεση Μαραγάλ. Τον ευχαριστώ για την τεράστια δουλειά που έκανε για ένα στρατηγική σημασίας και περίπλοκο θέμα σύμφωνα με το άρθρο 155 και σε συνεργασία με την Επιτροπή ε, για την Απασχόληση μπορέσαμε λοιπόν παρά τον, τις 221 τροπολογίες προχωρήσαμε, βρήκαμε μια συνθετική πρόταση, καταλήξαμε σε μια συνθετική πρόταση. Να πω ότι η γνωμοδότηση της απασχόλησης είχε 42 προτάσεις από τις οποίες μόνο οι 12 θεωρούνται αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης και γι' αυτό δεν θα ψηφιστούν, αλλά είναι στο τέλος του κατάλογου των ψηφοφοριών. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω εκτός κι αν ο Μαραγάλ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος θα ήθελα να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε, δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε η Προεδρός μας. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω όλους και ιδιαίτερα τη Γραμματεία. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό γιατί στη Γραμματεία δούλεψαν πολύ και καλά. Ε, το θέμα αυτό, η έκθεση αυτή παρουσίαζε ένα υψηλό βαθμό περιπλοκότητας και σε επίπεδο τεχνικό συνεργασίας ανάμεσα στη δική μας Επιτροπή και την Επιτροπή Απασχόλησης. Και υπάρχουν θέματα συζητήσιμα σχετικά με τα όρια ανάμεσα στα αρμοδιότητες των δύο Επιτροπών πάντως νομίζω ότι η προσπάθεια που έγινε απέδωσε καρπούς ε, έχει ενσωματωθεί η γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης στην ε, βασική μας έκθεση η οποία εμείς την ξεκινήσαμε, την οποία εμείς ξεκινήσαμε, αποφύγαμε κάποιες μορφές επικάλυψης, κάποια επίπεδα βέβαια έτσι κερδίσαμε θα έλεγα το ευανάγνωστο της έκθεσης, τη συνοχή της που περιγράφει σωστά τις θέσεις μας, τα κριτήριά μας και τις προτάσεις μας. Η έκθεση αυτή, σύντομα λέγω πρόεδρο, ε, δεν είναι νομοθετική πρόταση, εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνουμε προτάσεις ε, μέσω της εκθέσεως αυτής αποστέλουμε ένα μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι μόνο την Επιτροπή αλλά τα κράτη-μέλη και τα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους εργαζομένους της Ευρώπης. Στην ουσία λέμε ότι η κατάρτιση και η δουλειά συνδέονται πάρα πολύ στενά. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στον τομέα της εκπαίδευσης, το, το πρόβλημα δεν είναι μόνο στον τομέα των εργασιακό, αλλά νομίζω ότι ε, συνδέονται άμεσα οι δύο αυτοί τομείς, αλλά πρέπει να εργαστούμε στους μηχανισμούς διασύνδεσης της εφιούς σύνδεσης ανάμεσα στους δύο τομείς έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα αυθεντικό, ένα ουσιαστικό σύστημα ευρωπαϊκό επαγγελματικής κατάρτισης το οποίο να γίνεται κατανοητό και να αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι μόνο θέμα λοιπόν θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στα σχολεία, δεν είναι μόνο θέμα επαγγελματική αυτήρα κατάρτισης, δεν είναι απλό θέμα οργάνωσης της αγοράς εργασίας. Η έκθεση αυτή προσπαθεί να υποδείξει τους δρόμους τους οποίους θα μπορούσε να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη επί τη βάση της κατανομής των αρμοδιοτήτων στον τομέα. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε ένα καλό μέσο έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε αυτές τις ε, όχι απλά καλές προθέσεις αλλά τις ευφυείς νομίζω προτάσεις να τις κάνουμε πραγματικότητα για όλους τους νέους στην Ευρώπη έτσι ώστε να γίνουμε όλοι πιο Ευρωπαίοι και κυρίως καλύτεροι Ευρωπαίοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για τη δεσμευσή του. Στέλνουμε ένα χειρό μήνυμα και σήμερα θα έχουμε και τη δυνατότητα να συζητήσουμε απευθείας με τον Επίτροπο. Οπότε έχει και πολιτική αξία ε, ως κατεύθυνση της Επιτροπής μας ε, για το θέμα. Λέμε ότι χρειάζεται περισσότερη, περισσότερη προσοχή από εμάς. Ας περάσουμε στην ψηφοφορία. Έχετε όλοι τα καρτελάκια μπορούμε να ξεκινήσουμε. Παράγραφος 1, συμβιβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχή, εγκρίνεται. Περνάμε στη σελίδα 4. 168 υπέρ, κατά. Συγγνώμη, χωρίς την ψηφοφορία. Λοιπόν, για το πρώτο κομμάτι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ας πάμε στην πρώτη 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παραγραφός 1 προφορική τροπολογία δική μου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κα... 40, να το ελέγξουμε λέτε η πλειοψηφία ήταν υπέρ ε. ωραία να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 39 υπέρ α, συγγνώμη άρχεται η ψηφοφορία λέει πρόεδρος πέρας ψηφοφορίας Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε, επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 41 εισηγητή υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παίρναμε στην 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική 2 ε, εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 στην επόμενη σελίδα. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 ή 55, έχει κάνει λάθος η ομιλήτρια, 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική 3, η συγκεκριτού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλε 7, στη σελίδα 9. Υπέρ, κατά, αποχές, να ξεκινήσουμε την... να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την έμπλεπτα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 31 ε, χωριστή ψηφοφορία με, από, λόγω των πρασίνων υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Για το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται εισηγητού 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλε 13 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην 86 στην επόμενη σελίδα τζαμπάσκι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 91. Τη Μαλτέζε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην έμπλε 14 στη σελίδα 16. Έμπλε 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλε 20 υπέρ κατά αποχές συγγνώμη, ε, σε τμήματα, χωριστή ψηφοφορία, πρώτο κομμάτι από τους πράσινους υπέρ, κατά αποχές εγκρινέται, δεύτερο κομμάτι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 8 εισηγή του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλε 28 στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλε 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές υπέρ ξανά κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 116 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία για την 116 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 117 συγγνώμη έχει αποσυρθεί 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ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 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλε 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 150 υπέρ ε, τμήματική ψηφοφορία, κατά τμήματα πράσινη στο πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ κατά αποχές ξανά να δούμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 164 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά 164 έρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας Ε, λοιπόν, απορρίπτεται 166 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 174 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 179 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 178 υπέρ, κατά αποχές επαλήθευση Άρχεται η ψηφοφορία για την 178. Πέρας ψηφοφορίας. Ήταν δικό μου λάθος μάλλον. Ε, Κάποιο ε, στο χέρι του κατά λάθο. Λοιπόν, εγκρίνεται. 177 υπέρ κατά αποχέ. Εγκρίνεται. 175 υπέρ κατά αποχέ. Απορρίπτεται. 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 180 εισηγητού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική όχι συγγνώμη 188 Λιμπάτσκα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 185 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην τροπολογία 199 στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 203 να ελέγξουμε, να επαληθεύσουμε συγγνώμη τη 201 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 203 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 202 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 215 υπέρ κατά κατά αποχές εγκρίνεται 218 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε έμπλε 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλε 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλη 22 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην τροπολογία 11 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έπλα α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, αιτιολογική σκέψη ε, B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ίσως αν να ελέγξουμε αιτιολογική σκέψη Β τροπολογία 16 άρχεται ψηφοφορία Κρασνοδιεύσκη πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, έμπλε β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ετυλογική σκέψη C 20 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε, να επαληθεύσουμε την 20 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 στην επόμενη σελίδα. Λιμπάτσκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 που προτείνει η ΕΜΠΛΕ και περνάμε στην τελική ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεσης ε, στο σύνολό τη με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 4 αποχές, μία ψήφος κατά συγχαρητήρια στον συνάδελφο Μαραγκάλ. Ε, συγχαρητήρια και στους Σκιώδης και ευχαριστούμε και τη Γραμματεία. Ας περάσουμε τώρα στην δεύτερη ψηφοφορία της κυρίας Τόμα, αλλά δεν την βλέπω μεταξύ μας για την απαλλαγή για το 2014. Η επί τη αρμόδια είναι η Επιτροπή Κόντ, όπως ξέρετε, κατετέθησαν 26 τροπολογίες. Αν και χωρίς την εισηγήτρια θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε με τη συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ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 is is, an error in my, my list. Υπάρχει ένα λάθος στο δικό μου κατάλογο, λέει η Πρόεδρος. Okay, okay, okay, but it's not the right... Uh, okay. Alors, we go to eight. Πηγαίνουμε λοιπόν στην 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 11 ή μάλλον 12, 12 Προφορική τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Α, έχει ζητηθεί κατά διαίρεση ψήφος εδώ. Πρώτο τμήμα της 14 But yet we have not any more uh vote. We can vote now. Sorry. Allora, we can vote uh if you if you like also so, but in any case we can open the vote. uh Λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 14 πρώτο τμήμα. That is adopted. Second part. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Η 15 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 5, υπέρ, 4 συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 30, ή μάλλον 23 διορθώνει η πρόεδρος. Πρώτο τμήμα Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 24, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 25, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 26, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, τέλος. 24 υπέρ, 2 αποχές και 4 κατά. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και τους σκιώδης. now, now we go to an important point of the... Πηγαίνουμε σε ένα σημαντικό τώρα σημείο. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Το σημείο 6 στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία. Πρόκειται για σημαντική έκθεση αναφέρεται στην στρατηγική 2020. Έχουμε να κάνουμε εδώ. We are working. Sorry. If you can speak out of the room, please. We are continue our work. Thank. Allora. Eh, Qui noi Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να ασχοληθούμε με κάποια από συγκεκριμένα θέματα, προτεραιότητες για μας. Γνωρίζετε ότι η προθεσμία είναι η 25η Φεβρουαρίου, 16η απογευματινή για την κατάθεση των τροπολογιών και αρχές Απριλίου η ψηφοφορία. Θα δώσω το λόγο τώρα στον εισηγητή για να μας παρουσιάσει την πρότασή του και μετά θα δώσω το λόγο στους Σκιώδης και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ξέρετε ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω για αυτή την έκθεση εν συντομία. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι κατά την εκπόνηση αυτής της έκθεσης ε, έλαβαν χώρα πολλές συναντήσεις, ειδικότερα με τη Γενική Διεύθυνση Παιδείας, με τους Ευρωπαϊκούς Πολιτιστικούς Οργανισμούς που ασχολούνται με την παιδεία. Συναντήσαμε διάφορους οργανισμούς, εμπειρογνώμονε και υπουργού ε, παιδείας. Προσπάθησα δηλαδή να συζητήσω με ευρία γκάμα ενδιαφερομένων μερών για την έκθεση αυτή. Η έκθεση αυτή λοιπόν πρέπει να πω Εντάξει, όπω είπα, δεν θα μιλήσω για τα πάντα εδώ, διότι είναι πολύ ευρύ θέμα η παιδεία. Η έκθεση αυτή λοιπόν περιλαμβάνει τρία βασικά ζητήματα. Στο πρώτο κομμάτι τη έκθεση, ε, εάν τη διαβάσατε και είδατε και τις τροπολογίες, ε, θα το αντιληφθήκατε. Ε, αναφερόμαστε στις πλατφόρμες, οργανωτικές δομές, ουσιαστικά μετά από τις αλλαγές που έγιναν ε, πέντε έτη ε, μείωση των εστιακών σημείων, ε, έτσι όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όλα αυτά υιοθετήθηκαν από όλους τους ενδιαφερομένους που καλέσαμε και εξέφρασαν μάλιστα και την ικανοποίησή τους. Γεννήθηκε έτσι μια νέα γενιά ομάδων εργασίας. Αυτό ζητάμε εμείς με αυτή την έκθεση αφενός ε, να διευρυνθεί η σύνθεση αυτών των ομάδων εργασίας σε σχέση με τις παλαιότερες ε, ώστε να μην συμμετέχουν μόνο οι υπάλληλοι των Υπουργείων να συμμετέχουν και άλλοι εμπειρογνώμονες πέραν αυτών. Επίσης θέλαμε να διασφαλίσουμε καλύτερο συντονισμό εντός των επιτροπών ε, που έχουν στα θέμα εργασίας τους την απασχόληση. Θέλαμε λοιπόν να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή των συστάσεων από τα διάφορα φόρα που εργάζονται υπό την αιγίδα αυτής της πλατφόρμας. Δυστυχώς ο συντονισμό δεν είναι πάντα εύκολο ε, και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό ζητάμε οι άτυποι κρατικοί φορεί να συνεργαστούν μεταξύ του για την καλύτερη εφαρμογή αυτών των πολιτικών. Επίση, ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα στο ρόλο τη οικογένεια ε, στην παιδεία και στην εκπαίδευση θα πρέπει να υπογραμμίσουμε πιστεύω αυτή την προσέγγιση που βασίζεται στο ρόλο της κοινότητας. Community based approach. Όλες οι μελέτες ε, δείχνουν πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος των γονέων για την ανάπτυξη του ατόμου, του παιδιού δηλαδή. Ε, ο ρόλος λοιπόν των γονιών είναι ε, κρίσιμης σημασία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχουν εντόνωτερη παρουσία οι γονεί και εντό των οργανισμών, ε, των διαφόρων δομών, των ομάδων εργασία που ασχολούνται με την εκπαίδευση και την παιδεία. Η εργασία λοιπόν αυτή τη πλατφόρμα ε, θα πρέπει να περιλαμβάνει και την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σχολείων και οικογενειών. Ένα άλλο κομμάτι, το δεύτερο της έκθεσης, αφορά την ε, εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Σε αυτό το δεύτερο κομμάτι εγώ υπογραμμίζω το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δώσει αρκετή προσοχή στην μορφή που θα πρέπει να έχουν τα τεστ, οι εξετάσεις ώστε να φέρνουν επαρκή αποτελέσματα. Συχνά αυτό οδηγεί σε υποβάθμιση του επίπεδου της γενικής παιδείας. Και έτσι χάνονται ορισμένες δεξιότητες. Εγώ θυμάμαι ότι στην εκθέση λέμε σαφώς πως ε, η παιδεία δεν πρέπει να προσαρμόζεται μόνο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας ε, πρέπει να δημιουργεί και σωστούς ε, πολίτες ε, με αίσθηση της ευθύνης, ευθύνης τους ως πολιτών. Επίσης να επενθυμίσουμε ότι υπάρχουν και στοιχεία που δείχνουν ότι και σε ορισμένες χώρες είναι υπερβολικά επικεντρωμένη στις ακαδημαϊκές αρχές η εκπαίδευση ε, μόνο σε αυτό και αυτό δημιουργεί κενά στις, ε, στις αγορές εργασίας αλλά και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης παρατηρείται αύξηση της ανεργίας μεταξύ των πτυχιούχων και αυτό λαμβάνουμε υπόψη εδώ. Επίσης πρέπει να υπογραμμιστεί ο ρόλος της διαδικασίας της Μπολόνια και να επιστήσω την προσοχή σας και σε αυτή την πτυχή. Εγώ είδα και τις γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών που ισχυρίζονται ότι η διαδικασία της Μπολόνια περιλαμβάνει και στοιχεία αρνητικά κατακαιρματισμό, τυποποίηση ορισμένων πρακτικών, ε, κάποια επιβολή ομοιομορφίας ε, εκ των ανώ που οδηγεί σε απώλεια ορισμένων στοιχείων. Συχνά ξέρετε στη συστηματική εφαρμογή ορισμένων ενιών που προερχόνται από το, κόσμο, από το χώρο της αγοράς εργασίας στον ακαδημαϊκό χώρο δεν είναι τόσο επιθυμητό αναφέρομαι τώρα στον έλεγχο και τα λοιπά τέλος πάντων τα πανεπιστήμια δεν είναι πολυεθνικές μια άλλη παρατήρηση αφορά την κινητικότητα και η κινητικότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως το Εράσμους είναι σημαντική. Πρέπει ωστόσο να υπογραμμίσουμε την ανάγκη πιο ποιοτικής προσέγγισης ε, της διαχείρισης αυτής της κινητικότητας των φοιτητών. Το τρίτο κομμάτι αυτής της έκθεσης τελώς αφορά ένα ζήτημα ε, ιδιαίτερα επίκαιρο τη μετανάστευση στον τομέα της παιδείας. Αναφέρομαι στο ότι η μετανάστευση δεν είναι μόνο από τρίτες χώρες, ε, είναι, ε, ε, συμβαίνει και μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Και εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία που υπογραμμίζουμε. Αναφερόμαστε στην κινητικότητα των διδασκόντων, σημαντική για την ανταλλαγή βελτιστών πρακτικών μεταξύ χωρών με μεγάλη εμπειρία και χωρών με μικρότερη εμπειρία διότι τίθεται το θέμα της ε, φτωχής εκπαίδευσης, φτωχής παιδείας σε ορισμένες χώρες, ε, ελλειπούς παιδείας. Ε, αυτές οι χώρες πρέπει να δεχτούν περισσότερους ε, μετανάστες ακαδημαϊκούς. Ε, αναφερόμαστε εδώ και στα παιδιά που, έχουν, που είναι παιδιά οικογενειών μεταναστών σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Τέλος, ένα ζήτημα που δεν έχει συζητηθεί επαρκώς μέχρι στιγμής είναι το ζήτημα της ε, διαφυγής ε, εγκεφάλων. Συχνά μας απασχολεί το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι σπουδαστέ και αργότερα και οι εργαζόμενοι λέμε λοιπόν συχνά ότι αυτή πρέπει να είναι κινητική. Αυτή η κινητικότητα έχει επιπτώσεις και στην κοινωνία, ιδίω δε στις χώρες της Νότιας Ευρώπης αλλά και πολύ στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη διότι πολλά ταλέντα χάνονται, φεύγουν δηλαδή από τις ε, πατρίδες τους. Πράγμα το οποίο αποφέρει πλονέκτημα στις χώρες τις οποίες εγκαθίστανται. Όμως για τις χώρες από τις οποίες απεχώρησαν βεβαίως οι επιπτώσεις είναι αρνητικές. Λοιπόν, εγώ θα αρκεστώ σε αυτά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή που χαρίσατε στα λόγια μου. Σας προτρέπω να διαβάσετε την έκθεσή μου και να συντάξετε τροπολογίες εφόσον επιθυμείτε. Και... Μόνο μια παράκληση έχω, δηλαδή με τις τροπολογίες σας να μην αμφισβητήσετε την λογική διάρθρωση της εκθέσεώς μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτή την πολύ σαφή παρουσίαση των τομέων προτεραιότητας. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Να δώσω το λόγο στους σκιώδεις ε, συναδέλφους πρώτα απ' όλα, ε, Σοϊντρόβα και Τσούκ, Μαραγκάλ και Τσουκής. Uh, for his Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για το εξαιρετικό κείμενο. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ε, όλα τα ευρήματα. Η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο την αγορά εργασίας. Αφορά τις διαφορές φάσεις των σπουδών και ε, πρέπει να γίνεται καλύτερη διαχείριση της συνεργασίας ε, και καλύτερο συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην έκθεση υπάρχουν ε, συγκεκριμένες προτάσεις, η προσέγγιση που βάσει της κοινότητας, υποστήριξη προς τους διδάσκοντες, συμπεριλαμβανομένης της οικογένεια επίση ε, μας ενδιαφέρει ο τομέας εκπαίδευση σε συνδυασμό με τη μετανάστευση και την πρόληψη τη ριζοσπαστικοποίηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι η προσέγγιση αυτή του εισηγητού είναι πολύ σημαντική και τον ευχαριστούμε. Έχω κάποιε αμφιβολίε. Αμφιβολίε για ορισμένε από τι ε, δηλώσει του σημείο 13 για του στόχου. Ε, είναι καλός ο στόχος αυτός ε, και δεν πρέπει να τον εγκαταλείψουμε αλλά φυσικά η ποιότητα της ε, ε, εκπαίδευσης είναι σημαντική, αλλά αν δούμε τα πιο ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο, παρατηρούμε ότι στι χώρε αυτέ το ποσοστό των τυχιούχων είναι άνω του 40%. Αντίθετα με αυτό που αναφέρεται εδώ στην έκθεση ότι θέλουμε να επιτύχουμε, ίσω θα πρέπει να παρακολουθούμε περισσότερο την ποιότητα των προγραμμάτων αυτών. Ναι, συμφωνώ, αλλά ο στόχο αυτό του 40% πιστεύω ε, πρέπει να μην εγκαταλειφθεί σε καμία περίπτωση. Ε, συμφωνώ με τα όσα λέει ο συγγετής του σημείου 16 για τη διαδικασία τη Μπολόνια. Δεν συμφωνώ. Φυσικά υπάρχουν κάποια θέματα ε, που μπορούν να βελτιωθούν, αλλά θεωρώ ότι ε, συμβάλλει η διαδικασία της Μπολόνια για την ανταλλαγή ε, γνώσεων ε, και πρακτικών έτσι όλοι οι φοιτητές εποφελούνται από τον κοινό ευρωπαϊκό χώρο πιστεύω τα βασικά συμπεράσματα της Επιτροπής μας τα βλέπουμε στην εκθέση της συναδέλφου Λιμπάτσκα που υιοθετήθηκε πέρυσι και εγώ θα υποβάλω τροπολογίες και προσδοκώ στη συνεργασία μου με τον εισηγητή, τον οποίο ευχαριστώ για την εκθεσή του. Ε, e Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κουρτσουκ. Ευχαριστώ τον κύριο για την εργασία του και βρίσκω καλή την λογική διάρθρωση της εκθέσεως του. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι με την εκπαίδευση και κατάρτιση πρώτα πρώτα αποσκοπούμε στο να αναπτυχθεί η προσωπικότητα των ατόμων και όχι μόνο να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας. Χρειάζεται να αναπτυχθούν κατάλληλες στρατηγικές εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις κατάλληλες επενδύσεις για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Τονίζω επίσης ότι θα πρέπει να αποδώσουμε προτεραιότητα στην ποιότητα. Πρέπει να αρχίζει από νωρίς η εκπαίδευση και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όλα τα εκπαιδευτικά μας συστήματα να ενισχυθεί η δημιουργικότητα, να αναπτυχθούν τα ενδιαφέροντα των νεαρών ατόμων και οι ικανότητες τους να βελτιωθεί η συνεργασία για το λόγο αυτό μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Αρχών. Αυτό είναι ουσιώδου σημασία για να μπορέσουν να ενταχθούν και μετανάστες και πρόσφυγες με διαρκή τρόπο στα εκπαιδευτικά συστήματα και να εξασφαλιστεί ώστε όσοι ήδη έχουν αποκτήσει προσόντα αυτά να μπορούν να αναγνωριστούν. Ο κ. Χουντής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή μας για την έκθεση γιατί ξέρω ότι κατέβαλε σοβαρή προσπάθεια, μας την περιέγραψε σε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει στρατηγική σημασία για την ευρωπαϊκή προοπτική. Όμως θέλω να πω ότι παρά την ειλικρινή προσπάθεια της έκθεσης ορισμένα φαινόμενα περιγράφονται με ατολμία, όχι τις πραγματικές τους διαστάσεις, αν θελήσει κανείς να κάνει αποτίμηση στο πού βρισκόμαστε σε αυτό το τομέα, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Εκπαίδευση. Ποιος ευθύνεται για την υποβάθμιση της εκπαίδευσης και ότι όλο το βάρος έχει μεταφερθεί στις απλές δεξιότητες, την κατάρτιση, με βάση μόνο τις επιταγές της αγοράς κατά την άποψή μου ευθύνεται η κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη αντίληψη. Αποτίμηση, κωδικοποίηση, έκφραση αυτής της αντίληψης είναι η πολιτική της Μπολόνια, στην οποία ασκείται η συνθήκη της Μπολόνια, στην οποία όντως ασκείται μια κριτική, αλλά και εδώ. Ε. Έτσι είναι τα πράγματα. Η συνθήκη της Μπολόνια ουσιαστικά είναι υπεύθυνη για τον κατακαιρματισμό και για την αποδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος στο όνομα αυτής της συνθήκης η μόνη σύγκληση και συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη που είδαμε να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια είναι η τάση για εμπορευματοποίηση και η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης. Οι σπουδές όπως το διαπιστώνει σε ένα βαθμό η έκθεση, ξαναλέω, μετατράπηκαν σε εκπαιδευτικά προϊόντα και η στέρεη επιστημονική γνώση σε σκόρπιες γνώσεις και πρόσκαιρη κατάρτιση. Επίσης, μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι αποτυχημένο. Είναι αποτυχημένα, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που λέγω, αυτά που λέγονται προγράμματα κινητικότητας. Το διαπιστώνει σε ένα βαθμό η έκθεση, διαπιστώνει ορισμένα πράγματα, συγκεντρώστε τις εμπειρίες σας και δείτε ότι ουσιαστικά αυτά τα προγράμματα κατάντησαν καταναλωτικά, να έχουν καταναλωτικό χαρακτήρα και να ενισχύουν στρεβλά πρότυπα απλήρωτης εργασίας χωρίς δικαιώματα εν γέννη και ολοκληρώνω στο διαπιστωτικό μέρος ε, πιστεύω ότι ουσιαστικά έχουμε μια συρρήκνωση στην ευρύτητα των γνώσεων και στην ακαδημαϊκή ελευθερία. Επιτρέψτε μου για λίγο, το είχα κάνει και στην πρώτη συζήτηση, να σας δώσω μια σύντομη εικόνα για την κατάσταση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, τη χώρα, από όπου προέρχομαι, όπου αυτά τα προγράμματα της λιτότητας έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουμε απολύσεις ή διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών, υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται έντονα στη χώρα μου και όχι μόνο, διαπιστώνεται και αυτό στην έκθεση, της χώρες δηλαδή της Νότιας Ευρώπης, αυτή η διαρροή των εγκεφάλων. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες γιατροί, μηχανικοί, αλλά και άλλοι επιστήμονες από την Ελλάδα φεύγουν και δεν σταματάει αυτή η ροή. Και ναι, θα τελειώσω για, να γίνει και, και το σχήμα λίγο κατανοητό γιατί λέω αυτά που λέω. Επειδή υπάρχει, υπήρχε δωρεάν εκπαίδευση στην Ελλάδα, οι σπουδές ήταν πιο εύκολε. Έβγαλε γιατρούς, έβγαλε μηχανικούς. Αποτέλεσμα είναι τώρα, βγαίνουν, δεν βρίσκουν δουλειά. Γιατί δεν βρίσκουν δουλειά, γιατί υπάρχει η πολιτική τη λιτότητα. Τι λένε λοιπόν οι Γερμανοί και άλλοι. Έχετε μεγάλα ελλείμματα εκτός των άλλων διότι δώσατε πολλά για την παιδεία. Όμως τα αποτελέσματα αυτής της εκπαιδευτικής πολιτικής, δηλαδή γιατροί και μηχανικοί, τα καρπούν τη Γερμανία και άλλοι. Αυτό είναι το αντιφατικό της όλης κατάστασης. Επειδή πιστεύω λοιπόν... Για να ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Επειδή πιστεύω ότι το μέλλον ενός επιστήμονα για το οποίο συζητάμε δεν μπορεί να είναι ο φαύλος κύκλος κατάρτιση, απασχόληση, ανεργία, επανακατάρτιση και ούτω καθεξής, νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε τουλάχιστον στις διαπιστώσεις, τουλάχιστον στις προστάσεις, σε πιο ριζική αναθεώρηση της πολιτικής για την εκπαίδευση. Θα το κάνω αυτό με τις, συγγνώμη, θα το κάνω με τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ, τελείωσα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, αλλά πρέπει να τηρήσουμε το χρόνο μας, παρόλο που όπως είπα είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μαραγάλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή για την παρουσίαση της αρχικής πρότασής του. Νομίζω ότι είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης. Αυτό το σημείο εκκίνησης μας δίνει νομίζω μια αρκετά καλή εικόνα του πού βρισκόμαστε σήμερα, την κατάσταση των πραγμάτων γενικά. Μέσω των προτάσεων αυτών θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα, αν θα έλεγα να περιγράψουμε μια ευρωπαϊκή φιλοδοξία που μπορεί να υπάρχει στον τομέα αυτό. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει σε πάρα πολλές αλλαγές για να βελτιωθεί η κατάσταση και αυτή είναι και η δική μας ευθύνη. Εμείς επαναλαμβάνω στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν νομοθετούμε αλλά διατυπώνουμε στρατηγικές και ορίζουμε κάπως την πορεία των πραγμάτων όπως θα θέλαμε να είναι. Υπάρχει λοιπόν ένας χώρος ανωτά της εκπαίδευσης Υπάρχει ένας χώρος ανωτά εκπαίδευσης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως υπάρχει και ένα σχετικά ενοποιημένος χώρος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχουν δυνατότητες σύγκλησης, συνεργασίας στον τομέα της ποιότητας που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την εκπαίδευση στις διαφορετικές κοινωνίες όπως επίσης και υπογράμμιση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα δηλαδή τα εκπαιδευτικά συστήματα να είναι μεταξύ τους συνεργάσιμα και να μπορούν να δίνουν ευκαιρίες στους Ευρωπαίους φοιτητές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν όχι για λόγους απλά αρμοδιότητας αλλά για λόγους συμφέροντος πρέπει να προσπαθήσει να καθοδηγήσει την πορεία αυτή της σύγκλησης έτσι ώστε να βελτιωθούν τα ποιοτικά στοιχεία των εκπαιδευτικών συστημάτων και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όχι μόνο στα πανεπιστημιακά. Εμένα με ενδιαφέρει ε, όχι μόνο η πανεπιστημιακή εκπαίδευση αλλά και το μεγάλο, μεγάλος ρόλος τον οποίο παίζει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και νομίζω ότι θέτει τα θεμέλια, θέτει τις βάσεις για μια ουσιαστική ε, βελτίωση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε την κατάσταση της εκπαίδευσης ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω των εργασιών του ΟΣΑ και μέσω ε, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα αλλά χρειάζεται και μία προσπάθεια περιγραφής της κατάστασης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να υπάρξει ένα πραγματικά ευρωπαϊκό σύστημα περιγραφής της κατάστασης στην πρωτοβάθμια και ε, δευτεροβάθμια ιδιαίτερα στον τομέα της κατάρτισης των διδασκόντων στις δύο αυτές κατηγορίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα συστήματα εκπαίδευσης. Το σύστημα εκπαίδευσης σήμερα δεν είναι φυσικά κάτοχος της αποκλειστικότητας των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Το σχολείο εκπαιδεύει αλλά η κοινωνία κυρίως εκπαιδεύει και φυσικά και η οικογένεια εκπαιδεύει. Ε, υπάρχει όμως δυνατότητα σύγκλησης σε ορισμένους τομείς και θα πρέπει τα εκπαιδευτικά συστήματα να ερμηνεύσουν σωστά το πεδίο αυτό συνεργασίας. Τώρα, για την επαγγελματική κατάρτιση που ψηφίσαμε μια έκθεση, γι' αυτή θα πρέπει να διασφαλίσουμε την κινητικότητα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επαγγελματικής κατάρτισης, όπως επίσης και τα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά, θα πω από τους συναδέλφους να είναι σύντομοι. Hannibal. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ βέβαια πρώτα πρώτα τον εισηγητή, ο οποίος υπήρξε πολύ συνεργάσιμος και βοήθησε πολύ μέσα από μια πολύ θετική διαδικασία. Τον ευχαριστώ και πάλι. Όταν μιλούμε για εκπαίδευση, αντιμετωπίζουμε πάντα κατά κάποιο τρόπο την δυσκολία ότι η εκπαίδευση είναι βέβαια αρμοδιότητα των χωρών μελών. Το ξέρουμε αυτό όλες και όλοι. Η προσπάθειά μας λοιπόν να θεσπίσουμε ένα στρατηγικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύσκολο έργο. Νομίζω όμως ότι ο εισηγητής καλά τα κατάφερε. Έκανε μια προσπάθεια να το κάνει το έργο αυτό όσο γίνεται πιο ευρωπαϊκό. Εγώ συμφωνώ εν μέρη με τον τελευταίο συνάδελφο που μίλησε, ίσως όχι για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, αλλά πάντως για την εκπαίδευση των δασκάλων μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα για τους ε, δασκάλους, περισσότερες εκπαιδεύσεις να τους προσφέρουμε. Έχουν βέβαια το πρόγραμμα Έρασμος και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες και δεν βλέπω για ποιον λόγο άραγε να μην μπορούμε να βάλουμε μέσα σε αυτά, να εντάξουμε μέσα σε αυτά και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Κάτι που θα προσδώσει έναν πιο ε, έντονο ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Για τα πανεπιστήμια έχουμε κάνει προσπάθεια να τα ευθυγραμμίσουμε περισσότερο στις πανεπιστημιακές Ωστόσο αυτό υπήρξε και χρονοβόρο και δύσκολο. Για οτιδήποτε πάντως αφορά ανθρώπου μέχρι 18 χρονών, νομίζω εκεί μπορούμε να στοχεύσουμε περισσότερο στην εκπαίδευση των δασκάλων. Το κείμενο της εκθέσεως είναι καλό και πολύ μου άρεσε το τμήμα περί μετανάστευσης. Ωστόσο υπάρχουν δύο παραλήψεις. Δεν μιλούμε για πρόσβαση στην εκπαίδευση υπέρ εκείνων που έχουν λιγότερες δυνατότητες και έχουν για παράδειγμα μεταναστευτικό ιστορικό. Αυτό θα πρέπει να περάσει μέσα από τις τροπολογίες. Επίσης δεν λέει τίποτα για την ισότητα των φύλων. Εδώ στην Επιτροπή μας μιλούμε συχνά για ε, τις γυναίκες, για τα κορίτσια και εκεί χρειάζεται να κάνουμε μια προσπάθεια να τις εντάξουμε περισσότερο και να μπει και κάτι περισσότερο για το ευρωπαϊκό περιεχόμενο. Ε, αυτό. Κατά τα άλλα πάντως είναι καλή έκθεση. Ευχαριστούμε. Δίνω το λόγο στη συνάδελφο Τροπέλ που ζήτησε το λόγο και έχω άλλους δύο εγγεγραμμένους Evans και Λιμπάτσκα. Μοργάνο και Γραμματικάκης. Και έτσι θα κλείσουμε. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Okay. Ωραία, ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Κρασνοντεύσκη. Να αναφερθώ μόνο σε ένα σημείο κατά την ομιλία σας εστιαστήκατε στο ρόλο των οικογενειών και ότι χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία αυτών με τα σχολεία. Σε κάποιο βαθμό αυτό αληθεύει. Από την άλλη όμως γνωρίζουμε και πολλές μελέτες το αποδεικνύουν ότι για τα παιδιά και για τους μαθητές είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχουν δημόσια ιδρύματα στα νηπιαγωγεία, ε, στα σχολεία διότι ε, προσφέρουν ε, επιπλέον γνώση, προσανατολισμούς, δυνατότητες πρόσβασης και επαφής με την κοινωνία. Οπότε αυτό να γίνεται βάση δημοσίων ιδρυμάτων. και αυτό, αυτό βοηθάει και ιδιαίτερα και τα παιδιά των μεταναστών. Δεν είναι λοιπόν μόνο ζήτημα οικογενειών. Είναι τι κάνουν, τι μπορούν να κάνουν οι δημοσίοι φορείς μας και όταν μιλάμε και για εκπαίδευση των ε, διδασκόντων και αυτό είναι ζήτημα δημοσίων φορέων. Ευχαριστώ. E Ευχαριστούμε. Ε, Evans, παρακαλώ. Δεν είναι εδώ. Λιμπάτσκα, παρακαλώ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καθηγητά, Συμφωνώ με τους συναδέλφους μου που μίλησαν ήδη και που σας συνεχάρισαν σε ό,τι αφορά την προσέγγισή σας. Σε τρία πράγματα συμφωνούμε. Πρώτο, τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι αυτά που θα καθορίσουν πόσο καλή θα είναι η εκπαίδευση. Δεν πρέπει να είναι υπεύθυνα για το αν θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης ή όχι. Δεύτερο, για την ανάπτυξη των ανθρωπιστικών επιστημών. Πολύ σημαντικό και αυτό. Τρίτο, ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα είναι σαν την Ακαδημία του Πλάτωνος ε, στον πίνακα του Ραφαέλου, αυτό δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι μπορεί να επιτευχθεί. Εγώ έχω τρεις παρατηρήσεις ωστόσο. Μιλείτε για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και λέτε ότι αυτή δεν είναι επαρκής. Δεν είναι όμως μόνο η ποιότητα. Ζούμε σε μια διαφορετική πραγματικότητα πλέον. Χρησιμοποιούμε διαφορετικές τεχνολογίες επικοινωνίας. Έχουμε άλλες πηγές για την άντληση πληροφοριών. Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στη γνώση και στην πληροφορία. Ο δάσκαλος πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν τις διανοητικές τους ικανότητες Κύριε καθηγητά, θα μπορούσα να διαφωνήσω μαζί σας σε ό,τι αφορά την προσέγγιση. Μιλούμε για τα σφάλματα της διαδικασίας της Μπολόνια, έχει καλώς, αλλά η βασική της αρχή είναι σωστή και έχει βοηθήσει πολλές χώρες. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια για την διατήρηση της αυτονομίας να έχει η σχολή την ελευθερία διαμόρφωσης της εκπαίδευσης που παρέχει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφος κ. Μόργανο. Πολύ γρήγορα θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να μην είμαστε γενικόλογοι σε ένα τέτοιο έγγραφο οπότε πρέπει να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένες προτεραιότητες να υπογραμμίσω και εγώ ε, τις ελλείψεις όσον αφορά το ρόλο της ε, παιδικής ηλικίας αυτό το επιχείρημα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί επίσης συμφωνώ με τη συνάδελφο Λιμπάτσκα που υπενθύμησε το πόσο καλή είναι η διαδικασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, εφόσον θέλουμε την ελεύθερη κυκλοφορία να λειτουργεί ε, στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ευρώπη δεν, χρεια... δεν αρκεί να αναφερόμαστε απλά στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι ένα όριο. Εντάξει, όλα αυτά που οργανώνουμε αλλά εμεί ας μην, ας μην κάνουμε μια επιλογή που θα μας οδηγήσει προς τα πίσω και μετά δεν πρέπει να διαμαρτυρόμαστε αν υπάρχει διαφυγή εγκεφάλων. Ευχαριστώ. Και για να κλείσουμε ο κύριος Γραμματικάκης, παρακαλώ να είστε σύντομοι. Νομίζω ότι θα πω, δεν είναι πολύ πρωτότυπο να πω, ότι η έκθεση αυτή που κατά τη γνώμη μου θίγει πολύ σωστά πολλά θέματα είναι πολύ επίκαιρη αυτή τη στιγμή. Γιατί το πραγματικό πρόβλημα της Ευρώπης, το έχουμε πει πολλές φορές κυρία Πρόεδρε, ε, είναι η έλλειψη συνεκτικού πολιτισμού και συνεκτικής παιδείας. Εξού και η σημερινή κρίση. Τρεις παρατηρήσεις μόνο. Θα ήθελα την έκθεση πιο αυστηρή στο εξή θέμα ότι σιγά σιγά με την οικονομική κρίση και τις διάφορες λιτότητες που εφαρμόζονται σε ποικίλο βαθμό σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αποκλεισμός κυρίως από την ανωτάτη παιδεία, μεγάλων τμήματων του πληθυσμού, οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν τα σχετικά έξοδα. Εκεί θα ήθελα μεγαλύτερη έμφαση, θα το πω στις τροπολογίες. Η δεύτερο πάλι που θα ήθελα μεγαλύτερη ε, ε, έμφαση είναι ότι η παιδεία η σημερινή, πάλι κυρίως η ανωτάτη αλλά και οι κατώτερες βαθμίδες, προσανατολίζονται προς τις ανάγκες θα έλεγα της κοινωνίας η οποία κατευθύνεται από άλλους παράγοντες ενώ όπως ξέρετε όλοι σας η παιδεία πρέπει να έχει ένα γενικότερο περιεχόμενο και τρίτο θίγεται στην έκθεση αλλά πολύ λίγο η στροφή που υπάρχει τα τελευταία χρόνια προς μια ψηφιακή παιδεία που παίρνει πολλές φορές εκρηκτικές διαστάσεις έχει πολλά θετικά αλλά και μια πολύ μεγάλη απειλή ο ψηφιακός κόσμος όπως ξέρετε είναι και τα δύο Θέλει λοιπόν προσοχή η έκθεση, ξεκινάει σωστά και ελπίζω με τις τροπολογίες ότι θα ολοκληρωθεί σε ένα σημαντικό κείμενο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Να πω στην ε, συνάδελφο ότι πράγματι... Α, η κυρία Ward. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, υπήρξε μια σύγχυση. Είχα δει το όνομά σας, αλλά δεν είχα δει ότι είχατε επανέλθει. Σας ευχαριστώ, λέει η κυρία Ward. Θα συμφωνήσω με πολλά από αυτά τα οποία ακούστηκαν. Να υπογραμμίσω τρία πράγματα. Πρώτον, η εκπαίδευση στοχεύει στο μέλλον. Έχει σημασία να μην ξεχνάμε ότι συζητάμε για την δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, οπότε πρέπει να συνεργαστούμε έτσι ώστε να βελτιωθούν τα πράγματα και σε εμά αλλά και σε γειτονικέ χώρες. Απαιτείται λοιπόν να έχουμε μια προσπάθεια συνεκτικότητας ε, σε σχέση με ε, τα θέματα. Τώρα για την μη τυπική, μη παραδοσιακή μορφή εκπαίδευσης. Εγώ είμαι προϊόν αυτής της μορφής της εκπαίδευσης και πάρα πολλοί νέοι ε, το σύστημα τους έχει διώξει και στη δική μου χώρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα η εκπαιδευτική διαδικασία έχει γίνει πάρα πολύ ε, θα έλεγα πιεστική και αποτρέπει πάρα πολλούς νέους να την ολοκληρώσουν. Τώρα ο διαπολιτιστικός διάλογος, διαπολιτισμικός μάλλον διάλογος και οι μορφές εκπαίδευσης που μπορεί να δημιουργήσει εδώ θα ήθελα να παραπέμψω στην έκθεσή μου για τον διάλογο τον διαπολιτισμικό που είχε ψηφιστεί ε, πριν ένα μήνα στο Κοινοβούλιο σαν σημείο αναφορά. Τώρα επανέρχομαι στα σημεία 14 και 17 για τη στενότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για τη μείωση του θεματολογικού της πεδίου. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί δυσφορία όχι μόνο στους νέους, στους εκπαιδευόμενους, αλλά και στους εργοδότες. Εγώ είχα πάει σε μια εκδήλωση την οποία είχε οργανώσει η Siemens στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, και εκεί ε, ε, ο εκπρόσωπος της Siemens είπε ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία ακόμα και για αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με θέματα θετικά και πρακτικά. Έτσι λοιπόν οι τέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες πρέπει να είναι εκεί, πρέπει να είναι απαραίτητες χωρίς τη δημιουργικότητα, χωρίς τα οράματα, χωρίς την επιχειρηματικότητα, χωρίς την ικανότητα επίλυσης προγραμμάτων. Η επιστήμη, η καθαρή επιστήμη δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να καλύψει όλα τα προβλήματα. Τώρα, για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως είπε η προλαλή σας, ήδη πολλοί καθηγητές εργάζονται σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Έχουμε τα ψηφιακά μέσα, τα οποία είναι σε άμεση σχέση με το ευρωπαϊκό χαρακτηριστικό. Ja, ich hatte mich nochmal zu Wort gemeldet, auch wenn die Liste schon abgeschlossen war, weil einige Äußerungen mich schon dazu Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να πω κάτι και αναφέρομαι στο θέμα της οικογένειας Δεν είναι το θέμα να αντιτάξουμε την οικογένεια με τη δημόσια εκπαίδευση. Αντίθετα, αυτά πρέπει να προσεγγιστούν. Αυτά που λένε οι δάσκαλοι, οι ενώσεις των δασκάλων κλπ. λένε ξανά και ξανά ότι καμιά φορά η συνεργασία οικογένειας και σχολείου δεν πάει καλά. Και αυτό, η βελτίωσή της δηλαδή, μπορεί να βοηθήσει και στην αντιμετώπιση της ρίζοσπαστικοποίησης και αλλού. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερη επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Σε πολλούς τομείς αυτό δεν λειτουργεί καλά. Πρέπει να το τονίσουμε ιδιαίτερα στην έκθεση αυτή, ότι η οικογένεια δηλαδή παίζει ένα σημαντικό ρόλο και στο σχολείο και το σχολείο στην οικογένεια. Δηλαδή μπαίνει ο ένας στις, στα οικόπεδα του άλλου και είναι σωστό αυτό. Οι γονεί πρέπει να γνωρίζουν και ποια είναι η κατάσταση στο σχολείο. Και αυτή η μετάβαση ανάμεσα στον χρόνο της οικογένειας, στον χρόνο του σχολείου επίσης είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν συμβαίνει παντού. Και επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αντικατασταθεί ή να υποκατασταθεί καλύτερα η οικογένεια στο σχολείο ή το σχολείο στην οικογένεια. Καθόλου. και λέμε κιόλα ότι 40% των νέων έχουν πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευση ή τουλάχιστον αυτό πρέπει να είναι ο στόχος. Όχι, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι μπορούν να τα καταφέρουν πολύ καλά και εκτός ανώτατης εκπαίδευση. Εάν μπει αυτό ο στόχο του 40% και πάμε ντε και καλά να τον επιτύχουμε κατεβάζοντα το επίπεδο των σπουδών, αυτό θα ήταν λάθο. Ούτε είμαι βεβαία ότι αυτό το 40% των πτυχιούχων που υποτίθεται ότι θα είναι ο στόχο, θα είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι από άλλου που μπορεί να έχουν πάει σε επαγγελματικέ σχολές. Το πρόβλημα την Πολόνια δεν είναι λόγω τη δομή εκεί έχει απόλυτο δίκιο η Λιμπάσκα, δεν είναι η Μπολόνια καθε αυτήν, είναι η εφαρμογή τη Μπολόνια είναι η εφαρμογή της Μπολόνια στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εκεί ρόλο παίζει πώς διαμορφώνονται τα διδακτικά προγράμματα. Δεν έχει σημασία αν θα υπάρχει το προδίπλωμα και μετά το δίπλωμα ή όπως έχουν φτιάξει τώρα το μάστερ και το bachelor κτλ. Ο τρόπος είναι αδιάφορος. Δεν μπορώ να σας επιτρέψω περισσότερο χρόνο έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας τον αξιότιμο κύριο Πέτεριν και την κυρία Βανγκάλ της, ε, του Ευρωπαϊκού Οίκου Ιστορίας ή μάλλον του Οίκου Ευρωπαϊκής Ιστορίας και θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα πρώτα στις δύο τελευταίες παρεμβάσεις που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφενός και μετά πάλι στον εισηγητή. Αλλά παρακαλώ να είστε συντομότατοι. Ορίστε. Κύριε Έριξον, εσείς είστε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα είμαι συντομοτάτη. Ευχαριστώ πρώτα-πρώτα τον εισηγητή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει πολύ ικανοποιημένη με το σχέδιο εκθέσεως. Μας φαίνεται θαυμάσιο. Να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα, αν μου επιτρέπετε, όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα των ομάδων εργασίας, στην οποία αναφερθήκατε. Διευκρινίζω ότι οι ομάδες εργασίας ήδη έχουν ευρύτατη εκπροσώπηση, όχι μόνο από Υπουργεία κρατών μελών, έχουμε και εκπροσώπους από υποψήφιες χώρες του ΕΦΤΑ, της ΕΖΕΣ, της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθερών Συναλλαγών. Επίσης από τον ΟΣΑ, από οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ο ΣΕΝΤΕΦΟΠ, που ασχολείται με την επαγγελματική κατάρτιση, και από άλλα σχετικά. Και έχουμε και μια ανοιχτή επιλογή και έχουμε και ένα ανεπίσημο συντονιστικό όργανο. Γίνεται ένα είδος απογραφής. Σε, αυτό, σε αυτή την απογραφή δεν μας ε, υποστήριξε κανείς την ιδέα για νέα συντονιστικά όργανα. Έχουμε διεξαγάγει και πολλές ε, συζητήσεις ενδοϊπηρεσιακέ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συνεργασία μας με τους ενδιαφερόμενους φορείς stakeholder, έχουμε εξειδικευμένε συναντήσεις, συζητήσεις με τους ε, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ούτω Δηλαδή, νομίζω ότι η δομή είναι σωστή. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια που έγιναν για την εμπλοκή των γονέων, εμείς θεωρούμε ότι η προσέγγιση πρέπει να είναι συμπερικτική, συμπεριληπτική, δηλαδή να μπαίνουν μέσα και οι γονείς και οι τοπικές επιχειρήσεις, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, να αναμειγνύονται όλοι αυτοί στην εκπαίδευση. Έχουμε και ένα κατάλληλο εργαλείο το οποίο τονίζει ιδιαίτερα την ε, σημασία ε, και λέγεται Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για τα Σχολεία. Σε ό,τι αφορά την κινητικότητα έχουμε το νέο πρόγραμμα Έρασμος και εκεί γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας με καλύτερη προπαρασκευή, για παράδειγμα ε, στην ε, εκμάθηση των γλωσσών και να διευκρινίσω και ορισμένα πράγματα σχετικά με κάποια σχόλια που έγιναν στη διάρκεια της συζητήσεως να τονίσω την ανάγκη να είναι συγκρίσιμα τα επίπεδα μεταξύ των χωρών μελών σε όλα τα επίπεδα εκπαιδεύσεως. Έχουμε το European Qualifications Framework και εκεί υπάρχουν συγκρίσιμα επίπεδα και στα 8 επίπεδα της ε, εκπαίδευσης έχουμε και την ευρωπαϊκή αξιολόγηση, έχουμε τα λεγόμενα benchmark για παράδειγμα για να ε, εξετάζονται οι περιπτώσεις αυτών που δεν τα πάνε καλά στα μαθηματικά ή που εγκαταλείπουν πολύ νωρίς το σχολείο. Το ίδιο μιλήσατε και πολύ και συμφωνούμε και εμείς με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Έχουμε κάνει και πολλή δουλειά και στην ομάδα εργασία για τα σχολεία, ιδίως για την αρχική εκπαίδευση και την παραπέρα κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Ελπίζω ότι θα τα περισσότερα και σημαντικότερα. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν και πάρα πολύ ε, σύντομοι και ωστόσο πολύ περιεκτικοί. Θα δώσω το λόγο πάλι στον εισηγητή, κύριο Κρασνοϊγεύσκη. Το θέμα είναι να εκπληρωθούν οι προσδοκίες για γνώση έτσι τα πανεπιστήμια καλούνται να παίξουν τον ρόλο τους και έτσι θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν σωστά ε, η κοινωνία και η οικονομία ε, την λειτουργία των πανεπιστήμιων. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της παιδικής ηλικίας και εδώ τίθεται και το θέμα της αναπηρίας γενικά θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις στην ένταξη των ανθρώπων με αναπηρίες στα σχολεία στο σύνολο της Ευρώπης γιατί έχουμε διαφορετικά συστήματα με διαφορετικά επίπεδα αν θέλετε ένταξης. Λοιπόν, ο, ο, ο, ο κ. Κρασνοντεύσκη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Εγώ περιμένω τις δικές σας τροπολογίες και για ευχάριστες συζητήσεις στο μέλλον για να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές λύσεις. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ε, καλωσορίζω για μια ακόμη φορά την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για την Ευρωπαϊκή Ιστορία που είναι εδώ στην πλατεία, ξέρετε, ένα κτίριο που έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και επίσης και τον πρόεδρο του, τον κύριο ε, Hans Gert Bettering που ήταν και από τους ιδρυτές ε, του σχεδίου αυτού το 2007. Την κυρία Μπαγκάλ που είναι η team leader του ε, προγράμματος που θα μας πει σε ποια φάση βρισκόμαστε γιατί το 2016 προβλέπεται να ανοίξει ο οίκος της Ευρώπης ή το σπίτι της Ευρώπης συνδέεται το θέμα αυτό με τον πολιτισμό. Υπάρχει και μια επιστημονική επιτροπή ε, με επιστήμονες και ιστορικούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουμε με δύο συναδέλφους. οι οποίοι στην παρούσα φάση δεν είναι παρόντες. Και επίσης αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να πούμε ότι πρόκειται για μια διαδικασία η οποία ήταν αρκετά περίπλοκη. Βέβαια είναι φιλόδοξο το πρόγραμμα έτσι ώστε να δώσουμε μια πραγματική δυνατότητα αναγνώρισης της ιστορίας, των ιστοριών της Ευρώπης και της διαδικασίας ολοκλήρωσης από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τον 20ο αιώνα μέχρι σήμερα και η πολιτιστική πρόκληση που υπάρχει έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις ιστοριογραφικές παραδόσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την καταγραφή όχι μόνο των μεμονωμένων εθνικών ευρωπαϊκών ιστοριών αλλά του συνόλου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε συνεργασία και με άλλους παίκτες του τομέα του ιδίου αυτού τομέα όπως τα μουσεία, τα ερευνητικά Ινστιτούτα, τα πανεπιστήμια ε, όπως είπα προβλέπεται να ανοίξει τον Νοέμβριο. Θα είναι μια σημαντική προσφορά για τους επισκέπτες και θα είναι και ένας συμβολικός χώρος για το άνοιγμα του Ιδρύματος αυτού σε νέους επισκέπτες έτσι ώστε να γνωρίσουν περισσότερα, να εμπλακούν βαθύτερα Όλα αυτά είναι απαραίτητα και πρέπει να τα ενισχύσουμε. Γι' αυτό θεωρήσαμε χρήσιμο να παρουσιαστούν στην Επιτροπή Πολιτισμού, η οποία είναι από τους άμεσα ενδιαφερομένους στο συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα. Και ευχαριστώ εδώ και τον υπεύθυνο Γενικό Διευθυντή του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα κύριε Πέτερινγκ να σας δώσω το λόγο και μετά στην ε, επιμελήτρια που είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα αυτό έτσι ώστε μετά από όλες τις συζητήσεις που έγιναν να δούμε πώς εσείς βλέπετε την ουσία του εγχειρήματος αυτού, ποιες είναι οι προϋπτικές τις οποίες διανοίγετε και ποιες είναι οι δυσκολίες που σας περιμένουν και θα παρουσιάσουμε και μέσω PowerPoint ε, το πού βρισκόμαστε σήμερα και ποιο είναι το πρόγραμμα των εργασιών. Να πω επίσης ε, ότι ε, θα έλεγα εξ ονόματος όλων σας πριν από, από τα επίσημα εγγένεια να υπάρξει μία επίσκεψη της Επιτροπής μας και να μπορέσουμε μαζί σας να μοιραστούμε την εμπειρία σας. Θα σας δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο. Με, θα μου πείτε εσείς πόσο χρόνο θέλετε να μιλήσετε εσείς και πόσο η συνεργάτη σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Παραλίγο να πω αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κάτι που δεν μπορώ βέβαια, δεν επιτρέπεται πλέον να πω. Είμαι όμως επίτιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα κατά κάποιο τρόπο μπορώ να πω ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πάντως ε, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας και ιδίω διότι δίπλα μου είναι και η κυρία Βανγκάλ, ο Χάραλτ Ρέμερ πίσω συντονιστή στο εποπτικό Μα συμβούλιο, η κυρία Λαού και άλλε και άλλοι συναδελφοί και συνεργάτε. Άλλωστε βλέπω πολλά ε, πρόσωπα, άλλα βεβαίως είναι νέα, άλλα όμως τα γνωρίζω από τα χρόνια που ήμουν εδώ, 1979 έως 2014, 35 χρόνια, αν μου επιτρέπετε μια προσωπική παρατήρηση. Σε αυτά τα 35 χρόνια ποτέ δεν ήμουν μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού. Επομένως αυτό για μένα σήμερα είναι μια σημαντική εμπειρία. Θα ήθελα να πω ωστόσο ότι στα διάφορα καθήκοντα που εξετέλεσα είχα πάντοτε υπόψη μου και τιμούσα την εργασία σας. Υπάρχει και ένα παράδειγμα έμεσα σχετιζόμενο με τον Νίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Όσοι εξημών είστε παλαιότεροι και παλαιότερες ευρωβουλευτές θα θυμάστε την συζήτηση για τη δημοσιονομική προοπτική των ετών 2007 έως 2013. Τον Δεκέμβριο του 2005 στη διάσκεψη κορυφής οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν Τα κονδύλια για τον έρασμο που τον έχετε και σήμερα στην ημερήσια διαταξή σας ενέκριναν λοιπόν τα κονδύλια για τον έρασμο να περικόψουν κατά 3 δισεκατομμύρια τα κονδύλια αυτά. Είχα φρίξει τότε, ήμουν επικεφαλής τότε της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Βρετανών Συντηρητικών. Είχα πει λοιπόν και δεν θα το λησμονήσω ποτέ στη ζωή μου. Ήταν, μας είχαν προσκαλέσει αμέσως μετά από τα Χριστούγεννα ο τότε ε, αυστριακός καγκελάριος μας είχε καλέσει στην Hofburg στη Βιέννη γιατί αναλάμβανε την Προεδρία για να μιλήσουμε για τις δημοσιονομικές προοπτικές Πρόεδρος ήταν ο Ζώσεφ Μπορέλ έλαβα τον λόγο και είπα στον αυστριακό τότε καγκελάριο και μελλοντικό πρόεδρο της Ένωσης ότι εάν επιμείνετε στα 3 δισεκατομμύρια περικοπές η δική μας κοινοβουλευτική ομάδα θα πει όχι και είμαι βέβαιος ότι και οι άλλες πολιτικές ομάδες θα πούν το ίδιο πράγμα. Και αμέσως μετά μίλησε ο Μάρτιν Σούλτ που είναι σήμερα πρόεδρος του Κοινοβουλίου και είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και ο φιλελεύθερος Γκραμ Βότσον που σήμερα είναι ο Σερ Γκραμ και μάλιστα εκ, των, εκ μέρους των Πρασίνων είχε μιλήσει ο Ντανιέλ Κονμπέντιτ και ο Φρανσίς Βιούτς των Αριστερών. Όλοι μιλήσαμε μια φωνή. Ο Βόλφαν Σούσελ τα κατάφερε πολύ καλά έτσι ώστε να επανέλθουν τα 3 δισεκατομμύρια. Και αυτά επέτρεψαν σε εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές να συμμετάσχουν στις ανταλλαγές. Δεν επανελήφθη το σφάλμα αυτό, ευτυχώς, στην επόμενη δημοσιονομική, δημοσιονομική προοπτική 2014 έως 20. Αυτά ξέρετε εσείς καλύτερα. Έρχομαι τώρα στον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Πάντοτε εγώ είχα την επιθυμία να βλέπω ανθρώπους να συναντώνται, να ανταλλάσσουν απόψεις, να αλληλοκατανοούνται και να είναι διατεθειμένοι να πάρουν μια κοινή πορεία για το μέλλον. Αυτό είναι και το διανοητικό θεμέλιο στο οποίο βασίζεται η πρόταση για τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Ένας πρόεδρος κοινοβουλίου δεν έχει μόνο μια αντιπροσωπευτική αποστολή, ένα αντιπροσωπευτικό καθήκον. Πρέπει να δίνει και ουσία και εγώ απεφάσισα τα δυόμιση χρόνια, 2007 έως 2009 που ήμουν πρόεδρος του Κοινοβουλίου, να προτείνω ένα νέο έργο, τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Τα είχα πει και στις προγραμματικές μου τότε δηλώσεις του Φεβρουαρίου 2007 ότι θα φτιάξουμε έναν τόπο που θα μας θυμίζει το ευρωπαϊκό παρελθόν, τις τραγωδίες της, τις τραγωδίες του παρελθόντος αυτού, αλλά και τον τεράστιο πολιτισμό που απολαμβάνουμε στην Ευρώπη, ε, αλλά και τις τραγωδίες. Και ότι θα μας θυμίζει ότι τότε, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάποιοι άνδρες, τώρα θα έλεγα γυναίκες και άνδρες, σήμερα, διδάχθηκαν, εξήγαγαν τα συμπεράσματα από τις τραγικές συνέπειες των 55 εκατομμυρίων νεκρών. Έτσι λοιπόν ήθελα να είναι ένας τόπος της θύμησης αλλά και ένα τόπο που θα είναι στραμμένος προς το μέλλον. Με κύριο επίκεντρο την ιστορία του 20ου αιώνα, το βάρος του Εθνικού σοσιαλισμού και του σταλινισμού, αλλά μετά και την πορεία προς μια ευρωπαϊκή ενοποίηση και ότι αυτά θέλουμε να τα συνδέσουμε με μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ επιστημόνων, μεταξύ των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και ιδίως να προσελκύσουμε τους νέους και τις νέες. Τώρα εννέα χρόνια μετά όλα αυτά ηχούν σαν να είναι πολύ εύκολα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω όμως και τις συζητήσεις με την Επιτροπή Προϋπολογισμών στην οποία συμμετείχε πάντοτε και η κυρία Τρίπελ. Δεκαπέντε χρόνια ως Πρόεδρος Πολιτικής Ομάδας και ως Πρόεδρος του Κοινοβουλίου όταν διεξήγα συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έρχονταν σε μένα οι συνάδελφοι όταν όμω τέθηκε το θέμα του οίκου τη Ευρωπαϊκή Ιστορίας, εγώ ξεκίνησα να πάω να βρω του συναδέλφου και είδα πώ διαβιούν στα γραφεία του. και αυτό το λέω για να σα πείσω ότι αυτό ο οίκο τη Ευρωπαϊκή ιστορία είναι σημαντικό θέμα για μένα. Στην πολιτική μου σταδιοδρομία και δεν υπερβάλλω, τίποτε δεν υπήρξε τόσο δύσκολο ως εγχείρημα όσο αυτός ο οίκος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Δεν θέλω να σας παρουσιάσω όλε τι λεπτομέρειε πρόκειται πρωτίστως για έργο project, δηλαδή του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μου είπαν μετά, αγαπητοί πρόεδρε, γιατί να το αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή και το Συμβούλιο των Υπουργών. Αν είχαν μπει από την αρχή στη μέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, θα είχε καταστραφεί το έργο. Γιατί όπου λαλούν πολλά κοκόρια, ξέρετε. Όμως στο μέλλον θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα σημαντικό βήμα προόδου υπήρξε επίσης όταν ο τότε πρόεδρος Μπαρόσο με επιστολή του προς τον διάδοχό μου τον Πολωνό πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του έγραψε ότι θα συμμετάσχει στα τρέχοντα έξοδα, στις τρέχουσες δαπάνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν ο Ζέρζι Μπούζεκ έλαβε την επιστολή αυτή και την διένυμε, τότε είπαν και τα μέλη του Κοινοβουλίου που είναι στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, εντάξει, τότε λοιπόν δεχόμαστε και εμείς να χρηματοδοτήσουμε. Τώρα έχουν περάσει όπως σας εξήγησα 9 χρόνια. Η Σίλβια Κώστα θύμισε ότι τον Νοέμβρη αρχίζει ή μάλλον εγκαινιάζεται ο οίκος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Τώρα βέβαια δεν μπορεί κανείς απλώς να προτείνει ένα έργο και αυτό αμέσως οικοδομείται, χρειάζεται μια διαδικασία και αυτή η διαδικασία πρέπει να τηρείται. Υπήρξε πρώτα μια ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία συνέταξε πραγματογνωμοσύνη για το τι θα πρέπει υποτίθεται να είναι ο οίκος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Είπα εγώ θα είναι βασικά η ιστορία του 20ου αιώνα, αλλά ξεκινώντας από την Ελλάδα, Ρώμη, Αναγέννηση, Χριστιανισμός, όλα αυτά τα συστατικά στοιχεία της Ευρώπης. Και σε αυτό το Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων συμμετείχαν προσωπικότητες από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό την Προεδρία του καθηγητού Χίτερ που ήταν επικεφαλής του οίκου της γερμανικής ιστορίας με επίσης τον καθηγητή Μπόροντεϊ από τη Βαρσοβία που είναι σήμερα επικεφαλής του Συμβουλίου Επιστημόνων του Επιστημονικού Συμβουλίου που έχει συντάξει τα σχετικά με το περιεχόμενο το Επιστημονικό Συμβούλιο αντικαταστάθηκε μετά από ένα ε, συμβουλευτικό συνοδευτικό συμβούλιο, ε, επιστημονικό συμβούλιο όπου όπως είπα προεδρεύει τώρα ο κ. Μπόρο και συμμετέχουν προσωπικότητες όπως ο Νόρμαν Ντέιβις, ε, γνωστός ιστορικός από τη Μεγάλη Βρετανία και άλλες σημαντικές προσωπικότητες. Σημαντικό επίσης είναι να τονίσω ότι το Εποπτικό Συμβούλιο, η Board of Trustees αν θέλετε, είναι ευρύτατο πολιτικά, ώστε να μην γίνει τελικά το έργο αυτό μια, μιας μόνο πολιτικής παράταξης, αλλά να είναι ένα έργο το οποίο ε, να αφορά όλους. Θα σας αναφέρω τα ονόματα του Board of Trustees. Ο Μίγκελ Άρχελ Μαρτίνες Μαρτίνες εκπροσωπεί εμένα, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια Ευρωβουλευτής και μάλιστα και Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Ο αρμόδιος Επίτροπος Πολιτισμού, Τίμπο Ράφτσιτς, η πρόεδρό σας Σίλβια ε, είμαι βέβαιο ότι προφέρει καλύτερα τα ονόματα. Η Σίλβια Κώστα λοιπόν ω πρόεδρο τη Επιτροπή Πολιτισμού, ο Ζαν Ατουί, πρόεδρο τη Επιτροπή Προπολογισμών, ο κ. Σάουνταργκα, τον οποίο ακούσαμε ήδη, ο καθηγητή Μπόροτζέι, που αποκαθιστά και τον σύνδεσμο με το Επιστημονικό Συμβούλιο, ο υποκόμη Νταβινιού, πρώην επίτροπο, ο Ζεράρ Ονεστά, πρώην αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, ο Βόιτσε Κροσκόφσκι, πρώην Ευρωβουλευτής, Πίτερ Σάδελαν, πρώην Επίτροπος, Ρούντι Βερβόρτ, πρωθυπουργός της περιφέρειας Βρυξελών. Γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι χρειαζόταν πάντοτε να συντονιζόμαστε με τον Δήμο Βρυξελών και με την περιφέρεια Βρυξελών. Η Νταϊάννα Όλης, πρώην αντιπρόεδρο τη Ευρωβουλή. και ο Φρανσί Βιούρτς, πρώην πρόεδρο της Ενωτικής Έγινε η πρόταση λοιπόν όπως είπα τον Φλεβάριο του 2007 για το έργο και κλήθηκε πρώτα το Προεδρείο να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του την οποία έδωσε. Χρειάστηκε να βρούμε και το κτίριο. Ο Χάραλτ Ρέμερ λοιπόν, συντονιστής μας τώρα, τότε Γενικός Γραμματέας του Κοινοβουλίου, ο οποίος τα κατάφερε να νοικιάσουμε για 99 χρόνια το κτίριο Eastman Kodak. Δεν είναι ακριβώς καν ε, μίστοση, είναι περισσότερο... Είναι πάντως μια μακρόχρονη μίσθωση, όπως αυτή που ε, χρησιμοποιείται για γεωργικά κίνητα. Χρειάστηκε μετά και μια ομάδα η οποία να καθίσει να αναλογιστεί από την αρχή το πρόβλημα. Ε, με την Τάλια Βανγκάλ και με άλλους σημαντικότατους και ενθουσιώδεις συνεργάτες. Χρειαστήκαμε βέβαια και αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που έγινε πανευρωπαϊκά. Ένας χρόνος πέρασε μέχρι να ολοκληρωθούν όλα αυτά. Αν θυμούμε καλά, 28 αρχιτεκτονικά γραφεία συμμετείχαν και τελικώς κέρδισε το γραφείο Μπορέλ, το οποίο ε, ε, διαμόρφωσε εκ νέου το πτήπαλε στο Παρίσι. Άνθρωποι λοιπόν με μεγάλη γνώση. Η Τάλια Μπάουκ Βανγκάλ θα σας εξηγήσει τις λεπτομέρειες της διαρκούς εκθέσεως που θα καταλαμβάνει περίπου 4.000 τετραγωνικά μέτρα. Θα παρουσιάζεται εκεί η ιστορική πορεία του 20ου αιώνα αλλά και πριν από αυτόν και η ευρωπαϊκή απάντηση, η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Θέλουμε και θέλαμε βεβαίω να είναι και μια εμπειρία αυτή για τους επισκέπτες διότι θα πρέπει να μπορούν οι άνθρωποι ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτουν αλλά και με το επίπεδο της μόρφωσής τους αλλά και με το επίπεδο του ενδιαφέροντός τους να μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της ιστορίας ε, αφήνοντας ορισμένα τμήματα, επισκεπτόμενοι άλλα τμήματα η εμπειρία αυτή λοιπόν θα είναι και διαφορετική ανάλογα με το περιεχόμενο των ε, αιθουσών αλλά και την συγκέντρωση των ε, αντικειμένων καθώς και ο πρόεδρος πρόεδρος Πέτερινγκ ευχαριστεί τους διερμηνείς που κάνουν την προσπάθεια να αποδώσουν τα κάπως περίπλοκα λόγια του. Ε, θα τα λέω και λίγο πιο αργά, υπόσχεται ο πρόεδρος Πέτερινγκ για να δει τους διευκολύνω. Κυρίε και κύριοι, ο οίκος... Α, λίγο πιο αργά. Πιάνω, πιάνω, ναι. Ο οίκος της ευρωπαϊκής ιστορίας θα ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσιότητος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο οι ομάδες επισκεπτών για το Ευρωκοινοβούλιο και οι ομάδες επισκεπτών αποδέχτηκαν πολύ ευμενώς το Παρλαμεντάριουμ. Το Παρλαμεντάριουμ δεν ταυτίζεται με τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Το Παρλαμεντάριουμ εξηγεί τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναφέρεται μεν στον οίκο τη Ευρωπαϊκή Ιστορία, αυτό είναι απαραίτητο, αλλά ο οίκος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας ξεφεύγει από τα πλαίσια αυτά και περιλαμβάνει βεβαίως και τα άλλα θεσμικά όργανα και βεβαίως την κοινή μας ιστορία. Τώρα, κόστος. Η Τάνια Μπάουκ Βανγκάλ γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση των δαπάνων αυτών. Εγώ θα σας αναφέρω μονάχα το δημοσιονομικό πλαίσιο. Η αναδιαμόρφωση του κτηρίου Eastman μας κοστίζει 31 εκατομμύρια ευρώ. Για την ίδια την έκθεση προβλέπουμε 21,4 εκατομμύρια ευρώ και 3,75, 3.750.000 για την συλλογή. Το πώς διαμορφώνεται η συλλογή θα σας τα πει η Ιτάλια. Το σύνολο λοιπόν του έργου θα κοστίσει συνολικά 56 1,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Τα δε έξοδα λειτουργίας θα ανέρχονται σε 11,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Αν τώρα συγκρίνετε τα 56-7 εκατομμύρια ευρώ, κυρίε και κύριοι, βέβαια εκ πρώτη όψεω φαίνεται να είναι πολλά χρήματα αυτά. Αν δείτε όμω ότι το Rijksmuseum στο Άμστερνταμ κοστίζει πολλέ εκατοντάδε εκατομμύρια, το Μουσείο τη Ακρόπολη και είχαμε κοντά μας και τον διευθυντή του Μουσείου της Ακροπόλεως στην Κριτική Επιτροπή για την επιλογή του αρχιτεκτονικού γραφείου. Αυτό κόστισε πάνω από 100 εκατομμύρια. Για μένα λοιπόν είναι εκπληκτικό, αλλά αυτό προσπαθήσαμε κιόλας να κάνουμε, να μην επιτρέψουμε να αυξηθούν υπερβολικά οι δαπάνες. Να παραμείνει το κόστος λοιπόν σε κάποια πλαίσια και νομίζω το επιτύχαμε. Να πω ακόμη τελειώνοντας το εξής για τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις. η διήγηση, η αφήγηση μέσα από την πορεία της ιστορίας, θα σας τα εξηγήσει βεβαίως η Ιταλία Γκάουκ Βανγκάλ σε λίγο, σύμφωνα με τις βάσεις της συλλογής θα βασίζεται στην ιστορική πορεία. Αυτά βεβαίως θα τα εξηγήσει περισσότερο όπως είπα η κυρία Βανγκάλ τέλη του περασμένου έτους άρχισε η διαμόρφωση της εκθέσεως. Ήδη έχει προχωρήσει πολύ. Θα υπάρχει λοιπόν και μια έκθεση η οποία, ή μάλλον θα υπάρχουν εκθέσεις οι οποίες θα εναλλάσσονται και αυτό τώρα το πρώτο βήμα δηλαδή έχει σχέση με τη μετανάστευση, το μεταναστευτικό. Τα εγγένεια θα γίνουν τον Νοέμβρη φέτος. Πριν ολοκληρώσω την σύντομη αυτή παρουσίασή μου κυρίε και κύριοι ή αν μου επιτρέπετε να σας αποκαλώ συναδέλφους, επανέρχομαι στα κίνητρα για το φιλόδοξο αυτό έργο. Πιστεύω ότι πολλοί εξημών θα κατανοήσετε τα κίνητρα που με παρεκκίνησαν εμένα και άλλους να εργαστούμε για την υλοποίηση του έργου αυτού. Νομίζω ότι και μέσα στις παρούσες εξελίξεις που δεν θέλω να εμβαθύνω, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν βρέθηκε αντιμετωπή με τόσο βαθιά προβλήματα όπως τώρα. Είναι λοιπόν θεμελιώδες να επανέλθουμε, να ψάξουμε να βρούμε ξανά τις θεμελιώδεις αξίες μας για να αντλήσουμε από αυτές το θάρρος για να συνεχίσουμε το έργο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά τις θεμελιώδεις βάσεις, ένας από τους στόχους του οίκου Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα είναι να τονώσει, να βαθύνει τις γνώσεις των Ευρωπαίων για την κοινή τους ιστορία, οδηγώντας σε μια καλύτερη κατανόηση της κοινή πορείας. Τέλος, το ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει. Αν το καλοδούμε το πράγμα, είναι ένας πραγματικός θησαυρό και αν δεν τον διαφυλάξουμε τον θησαυρό και αν δεν επιφέρουμε τις διορθώσεις εκεί όπου πρέπει. Και βέβαια πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν και ιδίως πρέπει να ενισχυθεί και πάλι η ιδέα της αλληλεγγύης. Αν όμως η γενιά μας δεν επανέλθει στα θεμελιώδη, αν αφήσουμε να υποστεί ζημιά ή και να καταρρεύσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, θα είναι σαν το δέντρο εκείνο που έχει ζήσει εκατοντάδες χρόνια, το οποίο απορροφά το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και μας δίνει οξυγόνο, θα είναι σαν να το καταστρέφουμε, σαν να το αφήσουμε να ξεραθεί, στερώντας του τον αέρα. Γι' αυτό, βεβαίως και δεν είναι πανάκια αυτός ο οίκος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, είναι όμως ένα λιθαράκι σε μια κοινή πορεία να γνωρίσουμε την ιστορία μας χωρίς να εγκλωβιστούμε σε αυτήν. Η γνώση της ιστορίας πρέπει να είναι για μας το μέτρο για τη μελλοντική μας πορεία, το κοινό μας μέλλον. Αυτή είναι η βαθύτατη υπεποίθησή μου. Από όποια χώρα και αν προερχόμαστε, το μέλλον μας είναι κοινό. Παρόλες τις διαφωνίες, που βεβαίως είναι αναγκαίες για τη δημοκρατία, ας μην το λησμονούμε ποτέ και ας μην λησμονούμε ποτέ τις αξίες που μας συνδέουν. Και αυτό το στόχο έχει να εκφράσει το, ο οίκος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πατρίν για την παρουσίαση αυτή αλλά και για τα τελευταία σας λόγια θεωρώ και ελπίζω η πλειοψηφία των συναδέλφων να υποστηρίζουν ε, αυτό ε, το άνοιγμα του συμβολικού οίκου της ευρωπαϊκής ε, ιστορίας σε εποχές δύσκολες για την ταυτότητα, τη δημοκρατία και την πολιτική ταυτότητα της Ευρώπης. Εύχομαι λοιπόν να, να αναδείξει τη σπουδαιότητα όλων αυτών ε, το Ίδρυμα αυτό το δικό σας και για τις επόμενες γενιές ε, διηγούμενο με έναν διαφορετικό τρόπο την ιστορία, τα αίτια γέννησης της Ευρώπης. Ελπίζω λοιπόν ότι το έργο σας σε αυτό θα εξυπηρετήσει κυρίως να αποκαταστήσει τη σπουδαιότητα, τη σημασία, την κατεύθυνση του οικοδομήματος αυτού όπου ελεύθερα συμμετείχαν οι ευρωπαϊκοί λαοί Θεωρώ λοιπόν ότι θα, θεωρώ, λοιπόν, θα έχει τεράστια αξία. Να δώσω τώρα το λόγο για να μας παρουσιάσει σε εικόνες μέσω διαφανειών ε, το έργο αυτό, η κυρία ε, η οποία συμμετέχει και αυτή στις εργασίες οικοδόμησης του οίκου Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Να δούμε λοιπόν τι δουλειά έχει γίνει, τι δουλειά απομένει να γίνει αλλά να αποκτήσουμε και μια ολοκληρωμένη εικόνα με την παρουσίαση αυτή, μετά από την οποία θα μπορέσουν να πάρουν το λόγο και οι συνάδελφοι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού, όπως είπε ήδη ο κύριος ε, Πέτερινγκ, η δημιουργία του σπιτιού Ευρωπαϊκής ιστορίας ενός ε, σύγχρονου κέντρου ε, έκθεσης και τεκμηρίωσης βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο η ομάδα μας εργάζεται ε, για το έργο αυτό από τις αρχές του 2011 και βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην υπονομαζόμενη ενιολογική βάση, το θεμελιώδες έγγραφο του έργου όπου θεσπίζονται οι κανόνε για το σπίτι αυτό ήδη από το 2008. Τι θα είναι το σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας. Το μουσείο αυτό θα αποτελεί γέφυρα μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου ε, με πληροφορίες βασιζόμενες στις τελευταίες ιστοριογραφικές έρευνες ε, και με τη χρήση ενός ερμηνευτικού εργαλείου. Όλοι οι επισκέπτες λοιπόν, ανεξάρτητα από το πόσο γνωρίζουν ιστορία, θα, έχουν, θα αποκτούν μία ε, εμπειρία ε, από το μουσείο αυτό που θα αγγίζει όλες τις ε, αισθήσεις. Το, η μόνιμη έκθεση που θα ανοίξει τον Νοέμβριο, όπως ακούσαμε, θα προσφέρει στους επισκέπτες του τις ρίζες της Υπήρου θα επισημαίνει τις διαδικασίες και τα φαινόμενα του 19ου αιώνα, του ε, φαινόμενα εθνικισμού, τη βιομηχανική επανάσταση, τον κομμουνισμό, τον καπιταλισμό, την απεικιοκρατία κτλ. Και μετά θα εστιάζεται σε γεγονότα του 20ου αιώνα, συμπεριλαμβάνοντας την ευρωπαϊκή διαδικασία ολοκλήρωσης που διαμόρφωσε την Ευρώπη στην οποία κατοικούμε σήμερα. Η μόνιμη έκθεση του σπιτιού θα εστιάζεται, όπως είπα, σε ευρωπαϊκά φαινόμενα. Δεν αποτελεί το άθροισμα εθνικών ιστοριών. Αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί. Εστιαζόμαστε λοιπόν πραγματικά στην Ευρώπη στο σύνολό της. Σκοπός μας είναι στο σπίτι της ιστορίας οι επισκέπτες από όλη την Ευρώπη να αποκτούν μια ευκαιρία διαφόρων ερμηνεών βάσει επιμέρους γνώσεων και εμπειριών. Το σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα είναι ένας τόπος ε, πολυτομιακών συζητήσεων ε, για το παρελθόν της, ε, Ευρωπαϊκής, της Ευρώπης. Κάτι άλλο που κάνει μοναδικό αυτό το μουσείο είναι η πολυγλωσία του. Η μόνιμη έκθεση θα διατίθεται σε 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όσους περνούν συχνά από το παρκό Λεοπόλντο, ε, έχουν δει να μεταμορφώνεται το κτίριο μπροστά στα μάτια τους και είναι έτοιμο για να φιλοξενήσει εκατοντάδες αντικείμενα που μαζί και, άλλα, μαζί και με άλλα εκθέματα θα ε, αποτελούν το σύνολο της ε, έκθεσης. Η Γιάννη πρόσωψη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ωστόσο η εγκατάσταση της μόνιμης έκθεσης έχει ήδη ξεκινήσει. Τα πρώτα αντικείμενα, στοιχεία έχουν ήδη στερεωθεί στις οροφές. Εδώ βλέπετε τις φράσεις που θα χρησιμεύουν ως επισημάνσεις που θα καθοδηγούν τους επισκέπτες στις εκθέσεις. Οι επισημάνσεις αυτές θα αποτελούν κομμάτι μιας μεγάλης εγκατάστασης που εμείς ονομάσαμε ανεμοστρόβελο. Ήψους 27 μέτρων από κάτω μέχρι το πάνω μέρος της σκάλας και θα αποτελούν το έμβλημα του μουσείου. Θα αποτελείται από γράμματα και λέξεις που θα συμβολίζουν την εισαγωγή του αλφάβητου ως θεμελίου για την ιστορία και τη γνώση βάσει γραπτών εγγράφων. Θα γνωρίζετε ότι στη μυθολογία ο Κάδμος, ο αδερφός της ε, Ευρώπης, ε, έφερε το αλφάβητο στους αρχαίους Έλληνες ε, αναζητώντας την αδελφή του. Το σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας κατά πολλούς τρόπους είναι ένα μοναδικό μουσείο. Θέλει να αγγίξει εκατομμύρια επισκέπτες από την Ευρώπη που ενδεχομένως ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή ιστορία και την ευρωπαϊκή διαδικασία ολοκλήρωσης. Η μόνιμη έκθεση φιλοδοξεί να αποτελεί μόνιμη πηγή ερμηνείας του παρελθόντος της Ευρώπης. Θα προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους περί της κοινής ιστορίας της Ευρώπης και να διατηρούν ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης. Το σπίτι θέλει να εμπλουτίσει αυτές τις γνώσεις, να αφυπνίσει την περιέργεια, γιατί οι περίεργοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν να μάθουν περισσότερα και να εμβαθύνουν, να θέσει ερωτήματα. Πιστεύω ότι στο μουσείο μας ε, μάλλον ε, θα τίθενται περισσότερα ερωτήματα από ότι θα δίνονται απαντήσεις. Θέλει επίσης να δημιουργήσει ευκαιρίες ε, ε, προβληματισμού επί της ευρωπαϊκής ιστορίας. Θέλουμε το μουσείο μας να γίνει μια δεξαμενή ευρωπαϊκής μνήμης. Το λέω αυτό διότι αυτό αποτελεί τη βάση της εξέλιξης της ευρωπαϊκής κοινή συνείδησης. Η έννοια της κοινή μνήμης έχει καθορίσει τις ρίζες μας ε, και καθόρισε το πώς εμείς φτιάξαμε τις εκθέσεις αυτές με σκοπό την κριτική ανάλυση. Θα ανοίξει λοιπόν φέτος. Και σύμφωνα με το θεμελιώδες εγγραφό η ομάδα ακαδημαϊκών του έργου έχει ακολουθήσει τις κατευθύνσεις ώστε ο σχεδιασμός και η λειτουργία να αντικατοπτρίζουν ε, τις τελευταίες ε, ε, τάσεις ε, του μουσιολογικού σχεδιασμού. Θα υπάρχουν χιλιάδες σκηνογραφικά στοιχεία, αντικείμενα αναπαραγωγές ε, και διάφορες οπτικές απεικονίσεις ε, για την παρουσίαση της ιστορίας που θέλουμε να διηγηθούμε. Τα αλληλεπιδραστικά στοιχεία ε, όπως 14 ταινίε, ειδικά για τη μόνιμη έκθεση, θα συμβάλλουν σε μια εμπειρία που θα ικανοποιεί όλες τις αισθήσει. Η, παρότι η μόνιμη έκθεση βασίζεται στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ιστορία, προβλέπεται για κοινό άνω των 12 ετών, αλλά έχουμε δημιουργήσει και ένα τμήμα για οικογένειες με παιδιά μεταξύ 6 και 10 ετών. Η έκθεση παρουσιάζεται σε διάφορα ε, επίπεδα και ε, είναι πλήρως ε, περιγραφική. Αυτό σημαίνει ότι ο επισκέπτης θα μπορεί να κατανοήσει τα κύρια μηνύματα χωρίς να διαβάσει όλα τα κείμενα που υπάρχουν διαθέσιμα είτε μέσω μιας ταμπλέτας που παρέχεται είτε μέσω του έντυπου οδηγού. Και φυσικά όσοι θέλουν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο και να δουν πιο λεπτομερό στο περιεχόμενο θα τους παρέχουμε ακόμη περισσότερες πληροφορίες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι όπως το Parliamentarium, το σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα είναι δωρεάν. Η επιλογή της αφήγησης αυτής σε έναν μικρό χώρο ακολουθεί τρία βασικά κριτήρια. Καταρχάς επιλέγουμε τα θέματα τα οποία θα παρουσιαστούν μετά από τα ερωτηματικά που έχουν τεθεί. Ποια είναι τα κομβικά γεγονότα τα σχετικά ε, ε, με το σύνολο της Υπήρου. Ποιες είναι οι ιστορικές ευμηνείς και μνήμες που συνδέουν τις εθνικές και κοινωνικές ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διαφορετικό κάθε φορά τρόπο. Υιοθετώντα μια διευρωπαϊκή αντιμετώπιση, ο οίκος αυτός ε, κρατά πάντα ζωντανή την ευρωπαϊκή προοπτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα παραδείγματα δεν καλύπτουν επιμέρους τμήματα της Ευρώπης είναι δυνατόν ε, να συνδέσει κανείς με ερυθρά νήματα τα διάφορα τμήματα της έκθεσης και έτσι ο επισκέπτης ε, να ε, έρχεται σε επαφή και με τις διαδικασίες και με τις ρίζες και με τις υπάρχουσες, τους υπάρχοντες δεσμούς. Έχω κάποιες επιπλέον διαφάνειες του σχεδίασης της εκθέσεως έτσι ώστε να πάρετε μια εικόνα. Καταρχάς οι διαφορετική τα διαφορετικά θέματα και οι ομάδες έχουν ε, ε, σχεδιαστεί με τρόπο έτσι ώστε να αποφεύγεται η μουσιακή κόπωση ε, και να κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψης. Υπόθηκε επίσης ότι ο οίκος της ευρωπαϊκής ιστορίας θα έπρεπε να έχει και την η δική του συλλογή, η ίδια συλλογή. Βλέπετε εδώ τα πρώτα ε, αντικείμενα τα οποία ε, ε, έχουν έλθει σε εμάς το 2012. Τότε είχαμε συνοδεύσει τους τρεις προέδρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Όσλο όταν πήρε η Ένωση το βραβείο Νόμπελ. Ε, τότε 140 αντικείμενα συγκεντρώθηκαν ε, και είχαν εκτεθεί γύρω από την αίθουσα τελετής για την επίδοση του βραβείου. Ε, ταυτόχρονα συλλέξαμε και αντικείμενα και για τις διαμαρτυρίες οι οποίες είχαν εξελιχθεί εκεί κατά της ε, λιτότητας, πάντα δηλαδή ε, κρατάμε μια πολλαπλή οπτική. Από τότε η συλλογή αυξάνεται συνεχώς με αντικείμενα υψηλής σημασίας τα οποία θα εκτεθούν στη μόνιμη, στο μόνιμο εκθεσιακό χώρο. Θα υπάρξουν άνω ε, των χιλίων αντικειμένων τρισδιαστάτων, βέβαια δεν έχουμε τόσο μεγάλο χώρο, ε, το 2013 επισκεφτήκαμε 300 μουσεία στην Ευρώπη και πάρα πολλά αντικείμενα τα οποία ήταν κρυμμένα στις αποθήκες των μουσείων γιατί ξέρετε ότι από τα αποθέματα των μουσείων επιδεικνύονται σε μόνιμη βάση περίπου το 15 με 20%. Συνεπώς λοιπόν ε, έχουμε τεράστιους θησαυρού στα μουσεία της Ευρώπης. Τα αντικείμενα τα οποία συλλέγουμε λοιπόν θα φτάσουν τις 3.000. Δεν προέρχεται μόνο από μουσεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως βλέπετε εμείς στοχεύουμε και στην απόκτηση ε, προσέκθεση αντικειμένων και από χώρες ευρωπαϊκές εκτός Ένωσης. Ακολουθούμε μια θα έλεγα πολύ πρωτότυπη διαδικασία στην μουσιακή ιστορία. Πρέπει να υπογράψουμε τις συμβάσεις ενοικίασης, ε, ιδανισμού καλύτερα, για όλα αυτά τα αντικείμενα είναι μια διαδικασία περίπλοκη και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας θα ήταν δύσκολο να φτιάξουμε ε, τον οίκο της Ευρώπης χωρίς ε, την συνεργασία γενικών διευθύνσεων των οργάνων και κυρίως του Κοινοβουλίου, της ίνλο, της ε, ΣΕΙΦ που μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε το επίπεδο ασφαλείας, την DGI Tech για τα θέματα της ηλεκτρονικής και θέματα γενικά πληροφορικής, πρέπει να αναφέρουμε επίσης και την συνεργασία και με τους συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης για τη μετάφραση. Συνεργαζόμαστε για πάνω από δύο χρόνια. Η μετάφραση όλων αυτών των εγγράφων δεν είναι μια εύκολη διαδικασία γιατί κάθε κείμενο περνά από ε, σωστό έλεγχο για τη διασφάλιση της σωστής ποιότητας. Τα κείμενα είναι το 15% της εκθέσεως συνολικά, είναι τεράστια η προσπάθεια. Να πω επίσης ότι ήδη έχουμε μεταφράσει 2.500 ετικέτες σημάνσεις ε, ε, εκθεμάτων ε, που είναι απαραίτητα για να σημασιοδοτηθούν τα αντικείμενα αυτά. Σας έδωσα λοιπόν κάποια παραδείγματα έτσι ώστε να σας εντάξω ακριβώς μέσα σε μια εικόνα γενικότερη της προσπάθειας την οποία κάνουμε για να ανοίξει η έκθεση πλέον τον μήνα Νοέμβριο. Ο οίκος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας δεν είναι μόνο μία μόνιμη έκθεση και μία προσωρινή έκθεση. Το Προεδρείο υιοθέτησε ένα σημείωμα και με άλλες δραστηριότητες ε, εξ αρχής όπως ε, ε, η πολιτική επικοινωνίας, η, μια καφετέρια και άλλα επιμέρους θέματα αρκετές λεπτομέρειες. Προετοιμάζουμε επίσης και ηλεκτρονικά προγράμματα μάθησης για καθηγητές, δασκάλους, μαθητές, φοιτητές έτσι ώστε να γίνουμε και χώρο συζήτησης και έτσι προγραμματίζονται ήδη πάρα, πολλά, πάρα πολλές συναντήσεις. Θέλουμε να υπάρξει δυνατότητα επίσης ε, ε, ε, για ενδιαφέρουσες μορφές δημοσιεύσεων Ήδη ε, προσπαθούμε να προχωρήσουμε στη σύναψη εταιρικών ε, συμφωνιών και σχέσεων με διαφορετικού τύπου οργανώσεις ε, στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Αν συγκρίνω την προσπάθειά μας με τον δρόμο, εμείς φτάσαμε στα 26 περίπου, στο 26ο χιλιόμετρο ε, και πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε όπως ο μαραθρονοδρόμος το, ε, το επιθυμητό αποτέλεσμα στον σωστό, στον εύθετο χρόνο. Το Νοέμβριο θα σας δώσουμε ένα μουσείο χρήσιμο για όλους και έναν χώρο συζήτησης και έναν χώρο αντιπαράθεσης. Σας ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος Κώστα, νομίζω ότι άξιζε η παρουσίασή σας, ήταν πιστική θα έλεγα έχει υπάρξει ε, εντατική προσπάθεια να ξεπεραστούν οι δυσκολίες για ένα περίπλοκο θέμα μόνο και μόνο η επιλογή ε, θα έλεγα των ε, συμβολικών αντικειμένων εκθεμάτων είναι πάρα πολύ δύσκολο όπως επίσης και η συλλογή των τεκμηρίων και των ιστοριογραφικών τεκμηρίων ε, και η έκθεσή τους ε, είναι ένα θέμα που θα παραμείνει ανοιχτό γιατί παράλληλα με τις συλλογές, τα εκθέματα, τις εκθέσεις απαιτείται ε, μεγάλη παρουσία και στο διαδίκτυο και νομίζω ότι θα μπορέσετε να οργανώσετε και πάρα πολλές συζητήσεις πολυφωνικού πάντα τύπου όχι μόνο με εμπειρογνώμονες αλλά και με απλούς πολίτες. Θα δώσω το λόγο τώρα σε συναδέλφους που έχουν ζητήσει να μιλήσουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ και την δόκτορα Λαούς, όπως επίσης και όλους τους συνεργάτες της το γεγονός είναι ότι το Κοινοβούλιο έχει την αιγίδα, θα υπό την αιγίδα του, το σύνολο της πρωτοβουλίας αυτής, Νιούελ, Τρούπελ, Σβέρ και Μαραγκάλ. Δεν ξέρω αν έχουν ζητήσει και άλλοι συνάδελφοι το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Μια απλή ερώτηση. Να ρωτήσω τον κύριο Πέτρεγκ θα λέγατε το κόστος ε, και ο σχεδιασμός του σπιτιού Ευρωπαϊκής Ιστορίας θα βοηθήσουν ε, τα, την επιχειρηματολογία υπέρ της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν ναι με ποιο τρόπο. Εύχομαι να μην βάλετε μόνο αυτή η παράμετρος ε, υπόψη όπως τους τελευταίους μήνες αλλά είναι θεμητό το ερώτημα. Τρίπελ θα έρθει σε λίγο. Κύριος Σβέρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πέτριν για την παρουσίαση. Να ευχαριστήσω και την κυρία Βοκ Βανκάλ που μιλά σλοβένικα και τα καταλαβαίνει άψογα. Κύριε Πέτερινγκ, είστε ένας εξαίρετος Ευρωπαίος, αφοσιωμένος Ευρωπαίος και πρέπει να πω ότι μας έχετε λείψει τα τελευταία χρόνια στην ευρωπαϊκή πολιτική. Ε, τα τελευταία χρόνια τα οποία χαρακτηρίζονται από πολλές κρίσεις, πολλούς παράγοντες από σταθεροποίησης του οικοδομήματός μας. Πιθανότητα κανένας από μας δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ότι η κοινή ευρωπαϊκή ιστορία είναι κάτι ανύπαρκτο. Πιστεύω ότι υπάρχει μια γενικότερη Ευρώπη και πιστεύω ότι το σπίτι ευρωπαϊκής ιστορίας ε, θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή διάσταση όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικής αλλά και μεταξύ των πολιτών μας. Είμαι βέβαιος ότι η αίσθηση ότι είμαστε Ευρωπαίοι θα βοηθήσει να λειτουργήσουν καλύτερα και οι θεσμοί. Οι θεσμοί εστιάζονται και στον πολιτισμό φυσικά και είναι πολύ σημαντικό αυτός ο ευρωπαϊκός πολιτισμός να προσφερθεί στους πολίτες. Αυτή είναι η καλύτερη εγγύηση για να διατηρήσουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και στο μέλλον. Και πάλι σας ευχαριστώ που εγγύηστε αυτού του έργου και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που οι δικοί μου επισκέπτες οι οποίοι ε, ανέκαθεν επισκέπτονταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλέον θα μπορούν να επισκεφθούν και το σπίτι Ευρωπαϊκής Ιστορίας δωρεάν. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε κυρία Τρούπε. Σα um, σας ευχαριστώ Σίλβια, ευχαριστώ πολύ και για την ανάπτυξη του θέματος καθώς και για τις ομιλίες σα Όταν αρχίσαμε να συζητούμε την ιδέα του οίκου ευρωπαϊκής ιστορίας, μία σημαντική ιδέα ήταν να δείξουμε ότι δεν υπάρχει μοναχά μια ερμηνεία της ευρωπαϊκής ιστορίας, αλλά πλήρωνες. Γι' αυτό θα ήθελα να μάθω με ποιον τρόπο επιτυγχάνετε να παρουσιάσετε διαφορετικές ερμηνείες στους επισκέπτες και τις επισκέπτριες. Γιατί νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι ενδιαφέρον και σημαντική πρόκληση. Πώς να παρουσιαστούν δηλαδή οι διαφορετικές επιλογές σε ό,τι αφορά τις ερμηνείες και να προκληθεί και μια συζήτηση σχετικά με τις διαφορετικές ερμηνείες και το τι σημαίνουν αυτές έτσι ώστε να κατανοηθούν βαθύτερα οι συγκρούσεις και να προκύψει και μια βαθύτερη κατανόηση. Θα ήθελα να επεκταθείτε λίγο σε αυτά. Προετών είχαμε συζητήσει την ιδέα εφόσον δημιουργηθεί ο οίκος Ευρωπαϊκής Ιστορίας στις Βρυξέλλες είχαμε πει ότι θα ήταν καλό να δημιουργηθούν διασυνδέσεις και με άλλα μουσεία στην Ευρώπη, όπως το Μουσείο Κατοχής στη Ρήγα, Μουσείο στη Βουδαπέστη και άλλα σχετικά. Υπάρχουν αυτές οι διασυνδέσεις. Έχετε τη δυνατότητα να ε, τίνετε ας πούμε χείρα συνεργασία σε άλλα μουσεία στις χώρες μέλη και με ποιον τρόπο παρουσιάζεται η δυνατότητα αυτή στο μουσείο σας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαραγκάλ. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όσα ήθελα να πω, τα είπε μόλις η κυρία Τρίπελ, ε, κυρίως όσον αφορά τη διασύνδεση μεταξύ του Σπίτιου Ευρωπαϊκής Ιστορίας και της Ευρώπης και των πολιτών, των μουσείων, των χωρών, διότι πράγματι αποτελεί πηγή που θα εμπλουτίσει, θα εμπλουτίζει διαρκώς ε, πέραν από τις μόνιμες και τις προσωρινές εκθέσεις. Από ό,τι κατάλαβα οι εκθέσεις αυτές ε, θα μπορούσαν ε, να εξαχθούν κατά κάποιο τρόπο και να παρουσιαστούν σε άλλα μουσεία, αυτά που ανέφερε η κυρία Τρούπελ. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβαίνει και με άλλες δραστηριότητες και, και άλλες δραστηριότητες, που άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να ε, εκτεθούν στο δικό μας μουσείο. Δεν ξέρω αν πρέπει να το ονομάσουμε μουσείο. Είναι κάτι παραπάνω. Θα πρέπει να είναι μάλιστα κάτι παραπάνω από απλά μουσείο. Είναι το σπίτι της Ευρώπης. Ο οίκος της Ευρώπης. Ε, εφόσον δεν επικεντρώνεται μόνο σε εκθέσεις αλλά υπάρχουν πολλές αλήθειες, πολλές ερμηνείες όπως αυτές που καθόριζαν και εξακολουθούν να καθορίζουν την Ευρώπη γιατί η Ευρώπη είναι κάτι που ακόμη οικοδομείται, δεν είναι απλά ένα θέμα συζήτησης, είναι κάτι που ακόμη αποτελεί αντικείμενο έρευνας και εξήγησης. Έτσι λοιπόν... Η... Ξέρετε, όταν λέμε μόνιμη έκθεση, μόνιμη έκθεση σημαίνει ότι αυτό το σπίτι Ευρωπαϊκής Ιστορίας κατά κάποιο τρόπο θα αποτελεί προέκταση του κοινοβουλίου μας. Θα πρέπει δηλαδή και αυτό να είναι ένα κοινοβούλιο των Ευρωπαίων πολιτών ώστε να μπορούν να μπουν μέσα, να μιλήσουν, να ακούσουν, να ερευνήσουν ενεργά. Πιστεύω ότι αυτό το σπίτι ιστορίας θα πρέπει να είναι το καλύτερο φάρμακο, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι κάπως καταχρηστικά, φάρμακο κατά του ευρωσκεπτικισμού, κατά του Brexit. Εκεί ακριβώς ε, θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία να ξεκινά μία συζήτηση, μία συζήτηση με κάποιες αντιπαραθέσεις, αλλά που θα διασφαλίζει ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ανοιχτή, δημοκρατική, χωρίς αποκλεισμούς ε, αυτό ακριβώς που σημαίνει Ευρώπη, που σήμαινε Ευρώπη σε όλη την ιστορία μας, αλλά και που πρέπει να σημαίνει και στο μέλλον. Ευχαριστούμε κύριε Κρασνοδιεύσκη. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να εκφράσω τρεις ενδιασμούς που θα μεταφραστούν σε τρεις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα ήθελα να σας ρωτήσω, αγαπητή κυρία και αγαπητή κύριε, ε, Ποια έννοια εικόνα της Ευρώπης χρησιμοποιείτε όταν μιλάτε για ευρωπαϊκή ιστορία. Διότι εγώ είδα και τη Ρωσία στο χάρτη που μας δείξατε προλίγου. Η ερώτηση λοιπόν που προκύπτει από μένα είναι η εξή. Σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη γεωγραφική έννοια, όπου θα μιλήσετε και για τη ρωσική ιστορία. Διότι, ξέρετε, όταν είναι να μιλήσει κανείς για κομμουνισμό είναι δύσκολο να αποφύγει να μιλήσει για τη Ρωσία και μετά η Τουρκία θα συμπεριληφθεί και η τουρκική ιστορία δίπλα στη ρωσική στο μουσείο αυτό. Οπότε ξέρετε, ναι, όλοι λέμε ότι είμαστε ευρωπαϊστές, αλλά για ποια Ευρώπη μιλάμε. Γιατί η Ευρώπη υπήρχε και πριν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υπάρχει και πιθανότητα και μετά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν ενός πολιτικού έργου που δεν μπορεί να θεωρείς κανείς ότι θα υπάρχει για πάντα, ότι θα είναι αιώνιο. Τώρα, όταν μιλάμε για τη διήγηση της ευρωπαϊκής ιστορίας, ε, δεν μπορεί κανείς να αποφύγει τις θεολογικές πτυχές, δεν μπορεί να μην μιλήσει για το Θεό. Λέτε λοιπόν εσείς ότι πρόκειται για ένα πολιτικό έργο, ότι όλη η ιστορία του 20ου αιώνα αποτυπώνεται στο Ευρωπα... σε ένα πολιτικό οικοδόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά εγώ δεν είμαι και τόσο βέβαιος ίσως η ιστορία αυτή να μην έχει ολοκληρωθεί θα σας συμβούλευα λοιπόν να είστε λίγο επιφυλακτικοί λίγο προσεκτικοί ε, καθώς προτίθεστε να εξετάσετε την ιστορία από αυτή την άποψη αν αύριο το Ηνωμένο Βασίλειο βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μιλάμε πια για τον Ομόνο Βασίλειο στο μουσείο αυτό. Ξέρετε, είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Τρίτη ερώτηση μετά. Ευρωπαϊκή πρόπτικη. Μα τι σημαίνει αυτό. Τι, τι εννοείται με αυτή την έννοια. Γιατί η ευρωπαϊκή ιστορία, ξέρετε, είναι προϊόν εθνικών ιστοριών. Εθνικών ιστοριών που διασταυρώθηκαν με διάφορους τρόπους ε, ε, η ιστορία μεταξύ Πολωνίας, Γερμανίας, Πολωνίας, Ρωσίας Ε, ε, εμένα λοιπόν, επειδή με ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή ιστορία, έχω διαβάσει πολλά βιβλία, διαβάζω στα Ιταλικά την Ιταλική ιστορία, στα Αγγλικά την Αγγλική ιστορία, ε, για να δω τις διάφορες ε, οπτικές γωνίες, αλλά ευρωπαϊκή προοπτική, ευρωπαϊκή οπτική γωνία, τι σημαίνει. Τα βάζει όλα μέσα στο ίδιο καλάθι. Είναι πλάνη πιστεύω μια τέτοια προοπτική. Οπότε από αυτή την άποψη το μουσείο αυτό Υπάρχει περίπτωση από διδακτική άποψη να αποδειχθεί κάτι άγωνο. Υπάρχει κίνδυνος ε, ε, το ιστορικό, πολιτικό καθήκον να, να πάρει ε, όλο το χώρο από, τον καλλιτεχνικό, από την καλλιτεχνική πτυχή. Ενδιαφέροντα τόσα είπα, λένε οι συνάδελφοι και διάφορες απόψεις. Δίνω το λόγο στον κύριο Στρογεύσκη. Λοιπόν, ε, δέχομαι, πρέπει να παραδεχτώ ότι μου αρέσει αυτή η πρωτοβουλία. Αλλά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση αυτών που θα την υλοποιήσουν. Διότι πρόκειται για κάτι εξαιρετικά περίπλοκο. Όπως είπε ο καθηγητής ο κ. Κρασνοντεύσκη, είναι Ηράκλειο έργο δεδομένων των σημερινών συνθήκων στην Ευρώπη. Ουσιαστικά ε, πρέπει εσείς ε, να συνθέσετε το ευρωπαϊκό μοσαϊκό. Πρέπει να υπογραμμίσουμε κάποια στοιχεία. Θα ήθελα να μάθω σε ποιο βαθμό θα χρησιμοποιηθεί ο πολιτισμός ε, για την απεικόνιση της ευρωπαϊκής ιστορίας. Θα είναι πιο σημαντικός ο Γκούτεμπεργκ ή ο Σέξπιρ. Ο Σέξπιρ ή ο Ναπολέον. Ποιες δηλαδή ιστορικές προσωπικότητες ε, θα χρησιμοποιήσετε για να απεικονίσετε την ευρωπαϊκή ιστορία και ποια γεγονότα της ευρωπαϊκής ιστορίας θα απεικονίσετε ε, ε, για να τροφοδοτήσουμε ε, τους αυτούς μας με δύναμη και θάρρος και για να διδάξουμε τις επόμενες γενιές. Και επίσης πέραν του πολιτισμού και η πολιτική θα δείξει αυτή, αλλά τις κοινέ μας ρίζες. Ε, σκέφτομαι όμως επίσης και τον Μότζαρτ και το Σέξπιρ, τον Μπαχ. Επίσης δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σας για άλλο ένα λόγο δύο των απολέων φυσικά. Ε, είναι μια μορφή που αλλιώς τον βλέπουν στη Γερμανία, αλλιώς στην Αυστρία, αλλιώς στη Γαλλία και αλλιώς στον Ενωμένο Βασίλειο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα γεγονότα που υπήρξαν εμβληματικά ε, καθώς η Ευρώπη μεταβαλόταν. Εγώ υπήρξα στην Πολωνία υπουργό Πολιτισμού για πολλά χρόνια και δημιούργησα και το Κέντρο Αλληλεγγύης, άνοιξα το Μουσείο των Ευρωπαίων Εβραίων και ξέρω πόσο κοστίζουν όλα αυτά τα μουσεία. Για να είναι οικονομικά αποδοτικό ένα έργο αυτού του είδους, μπορείτε να μου πείτε πόσους επισκέπτες θα δέχεστε καθημερινά στο μουσείο αυτό ώστε να αποδίδει οικονομικά επαρκώς πόσοι θα μπορούν να μπουν να επισκεφθούν το μουσείο αυτό επίσης ένα τεχνικό ζήτημα πόσο χρόνο θέλει κανείς για να επισκεφθεί ολόκληρη την έκθεση φυσικά εξατάται από την ταχύτητα του κάθε επισκέπτη αλλά... αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο χρόνος είναι κάτι σημαντικό Κατά την άποψή σας, πόση ώρα θέλει κανείς για να περάσει από την έκθεση και να δει όλα τα εκθέματα. Δύο παρατηρήσεις τελικές να κάνω. Στο μεταξύ να ευχαριστήσω όλους για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όπως βλέπετε εκδηλώνεται τεράστιο ενδιαφέρον, φυσικά και πολλοί ενδιασμοί, ε, κάτι αναπόφευκτο όπως είπατε και εσείς. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις. Βάσει των όσων είπε ο συνάδελφος Κρασνεοτιεύσκη. δεδομένων των μεγάλων ε, ε, ιστορικών και πολιτιστικών κινημάτων που είδαμε στην Ευρώπη ε, πιστεύω και εγώ το θέμα των θρησκειών είναι σημαντικό υπήρξαν σημαντικές και ειδικότερα στον 20ο αιώνα η συμβολή για παράδειγμα ε, της ευρωπαϊκής κουλτούρας. Ε, είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα ο διαθρησκευτικός διάλογος, ε, η συμβολή όλων αυτών των φιλοσοφιών. Θεωρείτε θα ληφθούν υπόψη στις διαδικασίες γιατί μου φαίνεται δεν το είδα στο πρόγραμμα όταν είχε παρουσιαστεί. Πιστεύω ότι και αυτό είναι ένα παράγοντα που έχει πολλά να πει στην ευρωπαϊκή ιστορία. Το άλλο μου ερώτημα είναι πώ θα το διηγηθούμε στου μετανάστε. Έχουμε νέου πολίτε σήμερα στην Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν μια διήγηση για του Ευρωπαίου, αλλά και μια διήγηση που θα πρέπει ε, γλωσσικά, πολιτιστικά και από άψη συμμετοχή να λαμβάνει υπόψη και του μετανάστε. Αυτό ξέρετε για μα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα διότι πιστεύω ότι αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κάποιος που δεν θέλει να είναι απλά παθητικός φελεξονούμενος ε, θα κληθεί να συμμετάσχει. Ε, και μια τελευταία σκέψη. Και μετανάστες σημαίνει σημερινοί μετανάστες, αλλά μην ξεχνάμε και την ιστορία των ευρωπαϊκών μεταναστεύσεων. πρέπει να υπάρχει και αυτή η πτυχή, οι δύο μεγάλες ευρωπαϊκές μεταναστεύσεις του 20ου αιώνα, για παράδειγμα. Γιατί το λέω αυτό, διότι πολλές φορές παρατήρησα ότι οι ίδιοι πολίτες ε, που μεταναστεύουν στην Ευρώπη όταν βλέπουν ότι και η Ευρώπη υπήρξε πηγή μεταναστών, ότι έχει γνωρίσει αυτή την εμπειρία και αυτό δημιουργεί μια γέφυρα επαφής ε, με τους πολίτες αυτούς. Οπότε όλο αυτό το θέμα των μεγάλων γεωπολιτικών προοπτικών στην Ευρώπη που ζητήθηκε να δοθεί ε, προσοχή πιστεύω ότι αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα μπορεί αυτό να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες αλλά ε, πρέπει να υπάρχουν και κάποιες οπτικές γωνίες για τις διάφορες διαδικασίες που θα έχουν να πούν πολλά για το πώς οικοδομήθηκαν οι αξίες ε, της Ευρώπης. Ε, μπορείτε να μας το εξηγήσετε λοιπόν κάπως αυτό, να μας πείτε πώς θα δημιουργήσετε την επαφή μεταξύ των διαφόρων ερμηνεών της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ευχαριστώ. συγγνώμη, συνάδελφος Χιμένες. Συγγνώμη, εσείς είχατε σηκώσει πρώτο το χέρι. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν το είχαμε σημειώσει. Κύριε Χιμένες. Ευχαριστώ κύριε Πέτεριν για την προσπάθειά σας η οποία έχει σαν ένα στόχο ο οποίος έχει ένα στόχο μάλλον ο οποίος μας ενώνει και δεν μας διαιρεί προωθεί την ιδέα της ευρωπαϊκής ταυτότητας την οποία όλοι συμμεριζόμεθα θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν χώρες με περιοχές και αυτόνομες περιοχές με συγκεκριμένη ιστορική προέλευση αν θέλετε που χρησιμοποιούν όμως κάποιες φορές τις διαφορές αυτές ε, έτσι ώστε να προκαλούνται αντιπαραθέσεις και διαφοροποιήσεις που οδηγούν στην διέρεση των πολιτών. Πάντως υπάρχουν πολίτες που πιστεύουμε ότι υπάρχει αλήθεια και στα πλαίσια αυτά και οι διαφορετικές αλήθειες οι οποίες πολλές φορές δεν θα πρέπει να δημιουργούν διαφορές μεταξύ μας. Δεν μπορεί να υπάρξει συνένεση αν δεν γνωρίζουμε όμως το πεδίο, το πεδίο στο οποίο κινούμεθα, αυτό το οποίο συζητάμε. Έτσι μόνο η Ευρώπη θα μπορέσει να βρει μια κοινή ιστορία. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε λοιπόν πως το προϊόν της εργασίας του οίκου της Ευρώπης και η προώθηση της παιδαγωγικής της συνεργασίας μπορεί να βοηθήσει σε τομείς τους οποίους είναι απαραίτητη η βοήθεια αυτή πώς μπορεί να δημιουργηθούν λοιπόν εμπειρίες ε, ε, ενσωμάτωσης, εμπειρίες ολοκλήρωσης από τη μία χώρα στην άλλη. Και αυτή η αφήγηση, η ολοκληρωμένη συνενετική, η σφαιρική όπως την προτείνει ο οίκος της Ευρώπης με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει τμήμα της ιστορίας που διδάσκεται στα, ε, στις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε πολλά προβλήματα ξέρετε ε, ότι ε, μερικές φορές κάποιες αντιλήψεις ε, οδηγούν σε διαφορετικές περιγραφές των ίδιων ιστορικών συμβάντων από τα γαλλικά βιβλία ιστορίας σαν παράδειγμα με τα γερμανικά και επίσης θα πρέπει να μην αγνοήσουμε και την τοπική ιστορία, την ιστορία των μικρών τόπων των Δήμων και Κοινοτήτων και ελπίζω να προχωρήσει σωστά το σχέδιό σας. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ο πρόεδρος Πέτερινγκ, σας ευχαριστώ πολύ αγαπητή Σίλβια. Ευχαριστώ και εσάς αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι εφόσον μου επιτρέπετε να σας προσφωνώ με τον τρόπο αυτό είναι και το απλούστερο για μένα. Αν σας πω, κυρίες και κύριοι, μου φαίνεται κάπως σαν να μπαίνει μεγάλη απόσταση μεταξύ μας. Δεν επιμένω, αν δέχεστε όμως ε, θα μου κάνετε μεγάλη χαρά. Επιθυμώ τώρα να απαντήσω με τη σειρά των ερωτήσεων. Η Τάλια Βάουκ Φανγκάλεν ασφαλώς θα συμπληρώσει. Πρώτα, για ένα γενικό σχόλιο. Δεν υπάρχει και τίποτε που να είναι τέλειο. Πάντα θα υπάρχει κάτι που θα είναι ανοιχτό. Κάποιος θα βλέπει ότι κάτι λείπει. Αυτό οφείλεται στο ότι οι απόψεις μας διαφέρουν ακόμα και αν είμαστε στην ίδια πολιτική οικογένεια έχουμε διαφορετικές απόψεις. Αυτό σημαίνει ότι και στον οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας θα ε, προκύψουν διαφορετικές ερμηνείες, διαφορετικές ε, απόψεις. Ε, του ενός θα του λείπει το ένα, της άλλης θα της λείπει το άλλο. Τίποτα δεν μπορεί να είναι τέλειο. Όσο ζούμε θα πρέπει να διατηρούμε και την ικανότητα να μαθαίνουμε και να ανακαλύπτουμε. Και αν ανακαλύψουμε όταν θα είναι έτοιμος ο οίκος Ευρωπαϊκής Ιστορίας ότι λείπουν σημαντικά στοιχεία, να το πούμε για να μπορέσουν να συμπληρωθούν. Έχουμε άλλωστε και το στοιχείο των εναλλασσόμενων εκθέσεων για σημαντικά θέματα λοιπόν θα μπορούν τέτοιες εκθέσεις να τα λάβουν υπόψη. Πράγματα που λείπουν δηλαδή να τα συμπληρώσουν. Αυτό το λέω εισαγωγικά. Και τώρα θα έρθω κατά σειράν των ερωτήσεων. Για σας Άντριου. Επειδή έχετε το ωραίο αυτό όνομα Άντριου, δεν θα ρωτήσω αν είστε σκότος, αλλά γνωρίζω ότι ο Άγιος Ανδρέας είναι προστάτης της Σκοτίας και αυτό δείχνει την πολυφωνία του Ενωμένου Βασιλείου. Άντριο Λουά, ρωτήσατε αν αυτό ωφελεί τη Μεγάλη Βρετανία. Εγώ θα παρακαλέσω πρώτα-πρώτα τα μέσα, τα μίδια δηλαδή, στην χώρα σας, αλλά και σε άλλες χώρες βέβαια, να αντιμετωπίσουν αντικειμενικά τον οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Στην εφημερίδα Σαν προδιετίας γράφτηκε ένα άρθρο που έλεγε ότι ο οίκο Ευρωπαϊκή ιστορίας θα κόστιζε παραπάνω από 100 εκατομμύρια λίρε, μάλιστα, δηλαδή ακόμα περισσότερο από ευρώ. Και ότι δεν θα βάζει μέσα ούτε καν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και αυτό λέει η εφημερίδα Σαν ότι δεν θα βάζαμε μέσα τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο επειδή η ιδέα για τον οίκο ευρωπαϊκή ιστορία προερχόταν από ένα Γερμανό. Ε, αυτά δεν είναι αλήθειες και να τα διαβάζω στην εφημερίδα αυτό το πράγμα Γι' αυτό θα παρακαλέσω και στη Μεγάλη Βρετανία και οπουδήποτε αλλού να παρουσιάζει τα πράγματα στη βάση της αλήθειας. Ούτως ή άλλως θα προκύψει κάποια στιγμή η αλήθεια. Ούτως ή άλλως εφόσον κάποιος πει αναλήθειες αυτό κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Μεγάλη Βρετανία ελπίζω και εύχομαι μέσα από την παρουσίαση της Μεγάλης Βρετανίας και γνωρίζω ότι ειδικά στην περίπτωση τη Μεγάλη Βρετανία ε, αμφισβητείται ο οίκο Ευρωπαϊκή Ιστορία. Δικαίωμά σα είναι. Αν όμω έχετε καλή διάθεση, θα βρείτε ερμηνείε που σίγουρα θα είναι χρήσιμε και θετικέ για το Ενωμένο Βασίλειο, για το οποίο έχω πάρα πολύ μεγάλο θευμασμό διότι εκεί εσεί αναπτύξατε τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Και γι' αυτό επιθυμώ η Μεγάλη Βρετανία να παραμείνει στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και την Παρασκευή θα ληφθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις σχετικά. Ελπίζω ο Πρωθυπουργός σας Κάμερον και οι υπόλοιποι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μπορέσουν να βρουν τις κατάλληλες λύσεις ώστε να μπορέσει να παραμείνει η Μεγάλη Βρετανία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ωστόσο να ανακόψει και την παραπέρα πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται κάποια ισορροπία. Η δική μου συμβουλή, εγώ επί 7,5 χρόνια ηγήθηκα κοινοβουλευτικής ομάδα που περιλάμβανε ως μέλη και τους δικούς σας συντηρητικούς, Άντριου Λούχαν. Ίσως γι' αυτό να ασπρίσαν τα μαλλιά μου γρηγορότερα, αλλά μην ανησυχείτε, άσπρα θα τα μαλλιά μου και αν είχα μόνο δικούς μου μέσα στην κοινοβουλευτική μου ομάδα. Πάντα θα υπάρχουν διαφωνίες, πάντα θα υπάρχουν καυγάδες. Η σύσταση που μπορώ να δώσω στους Βρετανούς ό,τι αφορά την κρίση του για τον οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας θα είναι να πείτε ότι ακόμα και αν εμείς ως Βρετανοί δεν συμφωνούμε απόλυτα με την κοινή δράση της Ευρώπης και έχετε βέβαια και τα γνωστά σας opt-out παρόλα αυτά να στηρίξετε την ιδέα της ποικιλία, της πολυφωνίας με την ενιαία προσέγγιση του μεγάλου αυτού θησαυρού που είναι η δημοκρατία, η κοινοβουλευτική δημοκρατία, το δίκαιο και αυτά ξεπήρυσαν από τη δική σας χώρα σε μεγάλο βαθμό. αυτό είναι που ζητώ εγώ. Μπορεί να μας χωρίζουν πολλά πράγματα, αλλά ας εγγύψουμε στις αξίες που μας ενώνουν και που είναι η ελευθερία, η δημοκρατία, το δίκαιο και η ειρήνη. Και ελπίζω ότι στην βάση αυτών των αξιών θα αναπτυχθεί και θα διατηρηθεί η αλληλεγγύη οι αρχές μας, οι αξίες μας λοιπόν είναι αυτές που μας ενώνουν και ελπίζω και πιστεύω ότι αυτό θα βρει απήχηση και στην Μεγάλη Βρετανία. Θυμούμε και τον Winston Churchill που το 1946 στην βαρισίμαντη ομιλία του στην Ζηρίχη είχε τονίσει ποια πράγματα μας ενώνουν στην Ευρώπη. Για την κυρία Τρύπελ, Helga Τρύπελ, Μιλήσατε για τις επιμέρους ερμηνείες που είναι δυνατές. Έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει άλλωστε το απόλυτο της αλήθειας. Ο καθένας ερμηνεύει την αλήθεια διαφορετικά. Δέστε την έννοια απολυταρχισμός. Η Χάνα Άρεντ, μεγάλη Εβραία πολιτιολόγος, αποκατέστησε την ισότητα στις επιπτώσεις δύο απολυταρχικών καθεστώτων του κομμουνισμού με την έννοια του σταλινισμού και του εθνικού σοσιαλισμού. Είναι πολύ διαφορετικά τα ιδεολογικά θεμέλια των καθεστώτων αυτών και όμως οι εργαλειοθήκες που χρησιμοποίησαν τα πολιταρχικά αυτά καθεστώτα υπήρξαν ίδιες. Αυτό είπε η Χάννα Άρεντ. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να φτάσουμε σε πολύ διαφορετικές ερμηνείες. Σε ό,τι αφορά την διασύνδεση, και Τρίπελ, με άλλα μουσεία, αυτά θα σας τα εξηγήσει η Ιτάλια. Νομίζω είπε όμως πριν ότι 300 μουσεία έχουν συνεργαστεί μαζί μας. Μίλαν Σβέρ, σας ευχαριστώ πολύ για την ενθάρρυνση που μας δίνετε και λέτε ότι θα θέλατε πολύ να είμαι ακόμη παρόν και σε ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας αυτά. Προσπαθώ, ωστόσο είμαι και πρόεδρος του Ιδρύματος Κόνραντ Αντενάουερ και θα τοποθετηθώ και δημοσία για την διάσκεψη κορυφής της ε, Πέμπτης και Παρασκευής εδώ, ε, θα, θα τελεστεί εδώ στις Βρυξέλλες και να είστε βέβαιος ότι όσο ζω και όσο έχω τα μυαλά μου θα συνεχίσω να υπηρετώ το Ευρωπαϊκό Ιδεώδες και θα είμαι πάντα στο πλευρό σας. Και σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας για την πρόσβαση στον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας ότι θα πρέπει να είναι δωρεάν, σας παρακαλώ αυτό να το δηλώνετε και προς τα έξω και στο μέλλον, γιατί κάποιοι έχουν άλλες ιδέες. Πρώτα να ολοκληρωθεί η προσπάθεια και μετά θα το συζητήσουμε ξανά το θέμα. Η γνώμη μου πάντως είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσει να είναι δωρεάν η πρόσβαση στον οίκο της Ευρωπαϊκή Ιστορίας. Ωστόσο την απόφαση θα την λάβετε εσείς ως Ευρωβουλευτές και εγώ δεν επιθυμώ να αναμειχθώ. Για τον κύριο Μαραγάλο, ο οποίος απεχώρησε ωστόσο, παρόλα αυτά θα ήθελα να σχολιάσω βέβαια θα προτιμούσα να τον κάνω παρουσία του. Ήταν ε, σωστό αυτό που είπε, ότι πρέπει να δείξουμε την εξέλιξη, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, ότι δεν πρέπει να ε, ταχθούμε υπέρ μιας μοναδικής ερμηνείας της πραγματικότητας. Συμφωνώ. Εγώ αποφεύγω να χρησιμοποιήσω τον όρο μουσείο. Μπορεί βέβαια ε, να μιλήσει κανείς για μουσείο γιατί όντως η διαμόρφωση της συλλογή είναι παρόμοια με αυτήν ενός μουσείου. Αλλά το, ο οίκος Ευρωπαϊκής Ιστορίας είναι ανοιχτός προς το μέλλον δεν περιορίζεται μονάχα στην αναδίφηση και στην παρουσίαση του παρελθόντος. Εσείς κύριε Κρασνοντέψκι, αφού σας ευχαριστήσω πρώτα για τους διαφορετικούς τρόπους ενατένισης του οίκου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Γνωρίζω ότι στην Πολωνία διεξάγεται συζήτηση για γενικότερα την ερμηνεία της ιστορίας και γνωρίζω ότι ο καθηγητής Μποροτζέη, ικανότατος άνθρωπος, ο κύριος και επίσης έχουν διαφορετικές ερμηνείες για την ιστορία. Τι είναι η Ευρώπη τώρα, ορίζεται μόνο γεωγραφικά. Θα πω το εξής, στον πυρήνα βρίσκεται για μένα ε, το σύνολο των αξιών της Ευρώπης. Και σας είπα ποιες θεωρώ ότι είναι ε, ελευθερία, δημοκρατία, δίκαιο και ειρήνη. Εάν εκφραστεί αυτός ο πυρήνας νομίζω θα έχουμε ήδη πετύχει πολλά. Η συνάδελφός μου ε, Τάλια Βανγκάλ θα τα πει καλύτερα σε λίγο. Θα υπάρχει ένας μεγάλος χάρτης πάνω στον οποίο θα εμφανίζονται οπτικά οι διαδοχικές αλλαγές των συνόρων στην Ευρώπη. Και θα δούμε εκεί και τον ρόλο που παίζει η Ρωσία. Παρόλη την κριτική που ασκούμε στη Ρωσία επί του παρόντος δεν μπαίνω περισσότερο σε βάθος γιατί είναι πολύ πολιτική συζήτηση αυτή, δεν πρέπει ποτέ να βγάλουμε τη Ρωσία από το μυαλό μας ως ευρωπαϊκή χώρα, διότι το δυτικό μέρος της Ρωσίας είναι Ευρώπη. Έχω βεβαίως επικρίσεις για την Ρωσία επί του παρόντος, αλλά χρειάζεται να παραμείνει ανοιχτός ο διάλογος, διότι είναι αναγκαία η συμμετοχή της Ρωσίας και για την Τουρκία το ίδιο. Εγώ δεν είμαι υπέρ της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό ε, να διατηρήσουμε την συνεργασία με τους άμεσους αυτούς γειτονές μας. Αυτό που λέτε κύριε Κρασνοντεύσκη ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι αιωνία. Εγώ εύχομαι να διατηρηθεί στην ζωή πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να την ζήσουν και τα εγγόνια μου και τα δυσέγγονά μου διότι είναι σημαντικό ε, να διατηρηθεί η ειρήνη μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και λαών. Ας ευχηθούμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ενωμένη και δυνατή. Μιλήσατε ε, και μιλήσαμε για το Brexit, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Στην Ευρώπη υπάρχουν διαφορετικές αφηγήσεις βεβαίως Αλλιώς βλέπουν οι Γάλλοι τον Ναπολέοντα από ότι τον βλέπουν οι Γερμανοί ή οι Ιταλοί. Και βεβαίως αυτές οι θεωρήσεις παραμένουν ισχυρές και αυτές πρέπει να συζητηθούν και να συζητούνται. Και το γεγονός ότι μιλούμε για τα πράγματα αυτά, μίλησε κάποιος και για τα σχολικά εγχειρίδια. Ο καθηγητής Γιάκοψεν, ο καθηγητής μου λοιπόν ε, που παρακολούθησε το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο της Βιοβόνης, είχε συμμετάσχει και στην γερμανοπολωνική συζήτηση τότε και ήταν αρμόδιος για τα βιβλία της ιστορίας. Είναι λοιπόν θετική εξέλιξη το ότι τα πράγματα τα βλέπουμε αυτά και με διαφορετικό τρόπο. Για σας Μπόγκταν Αντζέι Ζορτογεύσκη θα σας πει για τους αριθμούς των επισκεπτών η Τάλια. Για το θέμα τώρα πολιτισμός και πολιτική. Η δική μου κατανόηση της ε, του πολιτισμού ε, περιλαμβάνει και την έννοια της πολιτικής, διότι η κοινή διαβίωση των ανθρώπων είναι και πολιτισμός και πολιτική. Και αν μιλήσουμε για μουσική, τέχνη και ούτω καθεξής, ναι μεν αυτό είναι πολιτισμός, αλλά παίζει ένα ρόλο εκεί και η πολιτική πτυχή. Αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ταυτόχρονα. Και άλλωστε οι μεγάλοι ποιητέ και στοχαστές της Πολωνίας και οποιασδήποτε άλλη χώρα, ευτυχώς και οι Γερμανοί έχουμε συνεισφέρει μεταξύ στοχαστών και ποιητών αν και κάναμε και μεγάλη ζημιά 33 μέχρι 1945 Ωστόσο θεωρώ ότι και η Γερμανία έχει συνεισφέρει στο πολιτιστικό γίγνεσθε της Ευρώπης. Μπορούμε να μιλήσουμε για τα πράγματα αυτά σήμερα που συναποτελούν τον μεγάλο ευρωπαϊκό θησαυρό. Για την Μαρία Τερέζα Γκίμινες Μπάρβατ, Χιμένες μάλλον, για την συμπερίληψη των περιφερειών και των επαρχιών. Ήταν απόλυτη πεποίθησή μας ότι πρέπει να αντισταθούμε στον πειρασμό να εξετάσουμε την Ευρώπη μοναχά από την σκοπιά των Βρυξελών ή του Στρασβούργου. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η Ευρώπη συνολικότερα που ξεπερνά τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε να εξετάσουμε μοναχά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη αρχίζει εκεί όπου καθένας έχει το σπιτικό του την οικογένειά του, τους φίλους του, όπου ενδεχομένως έχει γεννηθεί ή όπου έχει μετεγκατασταθεί, όπου, ε, όπου είναι η καρδιά του και το μυαλό του. Εμείς ε, στη Γερμανία λέμε για πατρίδα χρησιμοποιούμε και τη λέξη Heimat που ετυμολογικά προέρχεται από το σπίτι, home, heim. Αυτό λοιπόν είναι και η βάση, το θεμέλιο της Ευρώπης. Αν λοιπόν η Μεγάλη Βρετανία εγκαταλείψει την Ενωμένη Ευρώπη, υπάρχει μεγάλο κίνδυνο η ίδια η Μεγάλη Βρετανία να διασπαστεί. Γιατί μπορεί μετά η Σκοτία να σηκωθεί να φύγει από, το Ηνωμένο Βασίλειο για να επανενταχθεί στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν την πατρίδα μα, έχουμε τι χώρε μα. Εκεί εμείς λέμε πάλι για την πατρίδα το Fatherland, αλλού κάποιοι άλλοι λένε Motherland έχουμε την, ε, ο καθένας την δική του ηθαγένεια, αλλά έχουμε και την κοινή ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Και εγώ συχνά λέγω, και εδώ θα ολοκληρώσω σιγά σιγά, απευθυνόμενος και στην πρόεδρό σας κυρία Κώστα, όποιος βλέπει μοναχά την πατρίδα, δεν την υπερασπίζεται παρκώς. Και θυμίζω κάτι που είχε πει ο Φρανσό Μιτεράν και ήμουν πέντε μέτρα μακριά του όταν το έλεγε. Όποιος βάζει το δικό του έθνος πάνω από όλα τα άλλα γίνεται εθνικιστής και ο εθνικισμός καταλήγει στον πόλεμο. Γι' αυτό τα πράγματα αυτά σημαίνουν στην ουσία την ενότητα μέσα στην πολυφωνία. Και εδώ μπαίνουν και τα θέματα των περιφερειών που είπε η Σίλβια Κώστα και τα θέματα του μεταναστευτικού και αυτό είναι και το, ε, το νόημα του οίκου τη ευρωπαϊκή Ιστορίας ότι θέλουμε να προωθήσει τον διάλογο για την ιστορία μας, για το παρόν μας και για το μέλλον μας. Και αν το πετύχουμε αυτό νομίζω θα έχουμε πετύχει πολλά. Δεν θα πετύχουμε βέβαια όλα ίσως όσα θέλαμε. Βρίσκω ότι η διδασκαλία της ιστορίας είναι σημαντικότερη από ποτέ. Έχουμε το, το διαδίκτυο και όλες αυτές τις ε, μορφές επικοινωνίας που πάνε να υποκαταστήσουν πολλά πράγματα, χρειάζεται όμως να παραμείνουμε μέσα στα πλαίσια αυτής της ενατένισης. Ευχαριστώ και πάλι την Πρόεδρό σας. Δεν θα ξαναλάβω το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το έργο που επιτελείτε εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού Οι φίλοι μας στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, στην Επιτροπή Γεωργίας λαμβάνουν πολλά χρήματα, έχουν δηλαδή μεγάλους προϋπολογισμούς που μπορούν να χειριστούν. Αλλά είναι σημαντικό να κάνουμε κάθε τι το δυνατό να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολιτική, τα προγράμματα όπως ο Έρασμος, άλλα προγράμματα για τους νέους, να είναι ενισχυμένα και εξασφαλισμένα. Και σας βεβαιώ ότι θα αναλώσω κάθε δυνατή προσπάθεια και κάθε δύναμη για να προωθήσω όσο μπορώ από την θέση μου τα πράγματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη ε. συναρπαστική δουλειά που κάνετε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία σε όλους και σε κάθε ένα σας ξεχωριστά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Ευχαριστώ τον ε, κύριο Πρόεδρο για τις παρεμβάσεις του. Θα είμαι πολύ σύντομη, έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει πολύ χρόνος. Όλα τα μουσεία τα οποία αναφέρατε συνεργάζονται μαζί μας. Υπάρχουν άνω των 300 μουσείων που θα μας ε, δώσουν ε, εκθέματα και είναι η αρχή της συνεργασίας αυτή ε, κάποια από τα εκθέματα θα μας δοθούν για βραχυχρόνιες μισθώσεις, κάποια άλλα ε, ε, διάρκειες ε, μάλλον. Αλλά για πιο μακροχρόνιες έχουμε λοιπόν δίκτυα συνεργασίας, έχουμε συνεργασία να το πω αλλιώς επίσης με δίκτυα που ασχολούνται με την ευρωπαϊκή ιστορία. Τώρα για την ερμηνεία των εκθεμάτων. Ένα παράδειγμα ίσως λίγο προσωπικό. Το δεύτερο τμήμα του 20ου αιώνα είναι κάτι το οποίο αποτελεί φυσικά τις αμνήμες της δικής μου γενιάς και των νεότερων γενεών. Στη δική μου ομάδα είμαστε ιστορικοί από διαφορετικές χώρες και επί τη βάση των, των ιστοριογραφικών δεδομένων Έχουμε και τις προσωπικές μας εμπειρίες βέβαια και τα αντικείμενα, αλλά μάθαμε για την μόνιμη έκθεση ότι λόγω ακριβώς των εθνικών ε, ε, προγραμμάτων διδασκαλίας ιστορίας έχουμε περιορισμένες απόψεις ε, και βλέπουμε την ιστορία των άλλων εθνών με πολύ στενό τρόπο. Και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σαν παράδειγμα εμείς λέμε ότι ο πόλεμος αυτός ήταν ένα συνολικός πόλεμος και ο τρόμος ε, έφτασε σε επίπεδα τρόμου και φρίκης που δεν είχαμε ποτέ φτάσει στην Ευρώπη. Και προσπαθούμε παρόλα αυτά να υπογραμμίσουμε και τα φαινόμενα της αντίστασης και τα φαινόμενα της συνεργασίας με τους κατακτητές. Ε, βέβαια ένα Ιρλανδός Ευρωπαίος θα έχει μια δική του ερμηνεία από αυτόν ο οποίος προέρχεται από την Πολωνία. Επί τη βάση λοιπόν των, ε, ιστοριογραφικών δεδομένων και της μουσιακής, μουσιολογικής μάλλον επιστήμης δίδονται συγκεκριμένες ερμηνείες. Αυτά έχουμε κυρίως μάθει από τη διαδικασία αυτή η γνώση πολλές φορές είναι προσωπική, είναι ε, περιορισμένη, θα θέλαμε να τη διευρύνουμε και να περάσουμε σε διαδικασίες ε, οι οποίες ε, να απηχούν με τον ίδιο τρόπο σε πολλές ταυτόχρονα χώρες. δεν μιλάμε μόνο για ένα απλό μουσείο. Εγώ εργάζομαι σε μουσεία 36 χρόνια και έχω δει πάρα πολλές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις των σύγχρονων μουσείων. Δεν είναι χώροι εκθέσεων εδώ και 20 χρόνια περίπου. Είναι κέντρα τα οποία χρησιμοποιούν την ιστορία και αναφέρομαι στα μουσεία τα ιστορικά έτσι ώστε να έρχονται στην επικαιρότητα συζητήσεις για το παρόντε και το μέλλον. Νομίζω λοιπόν ότι έτσι θα πρέπει να λειτουργήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Δεν έχουμε μόνο την μόνιμη εκθέταση, ε, έκθεση, συγγνώμη, έχουμε και την προσωρινή έκθεση. Ξεκινάμε ε, τον Νοέμβριο με διάφορες ανταλλαγές που μας δίνουν την ευκαιρία να εμβαθύνουμε τις γνώσεις τις οποίες έχουμε ε, και για τα δεδομένα της μόνιμης έκθεσης στην οποία δεν μπορούμε να πάμε σε πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Έχουμε επίσης προγραμματίσει και μια περιοδεύουσα έκθεση η οποία είναι καρπός της συνεργασίας με πολλές άλλες χώρες. Δεν έχουμε μια τελειολογική θα έλεγα αντίληψη, έχουμε μια πολιτική αντίληψη αξιολόγησης δηλαδή των πολιτικών διαδικασιών που βρήκαν χώρο στο δικό μας μουσείο η, η ευρύτερη Ευρώπη, η μεγάλη Ευρώπη, η γεωγραφική Ευρώπη, ήδη ο μύθος της Ευρώπης δείχνει ότι η Ευρώπη ανέκαθεν ήταν ένα επίπεδο διαπολιτισμικών ανταλλαγών. Η Ευρώπη, Ευρώπα ποτέ δεν περιορίστηκε σε συγκεκριμένα όρια της Ευρωπαϊκής Υπήρου και μάλιστα μετά από και την έρευνα που κάναμε εντυπωσιαστήκαμε από το πόσο λίγοι Ευρωπαίοι γνωρίζουν τον μύθο της Ευρώπης. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά. Τώρα για τις προσωπικότητες υπάρχουν πολλές. Τώρα για τη μετανάστευση, για τους μετανάστες μάλλον. Έχουμε 6 ομάδες και 23 επιμέρους θέματα. Η Ευρώπη είναι προϊόν μετανάστευσης, δεν μπορούμε να μην το πούμε αυτό στο εισαγωγικό κεφάλαιο και στο έκτο κεφάλαιο λέμε εμείς ότι ήδη ε, περιλαμβάνονται στη συλλογή μας αντικείμενα μεταναστών από τη Μεσογειακή Λεκάνη από αυτούς που ήρθαν πέρυσι. Είναι λοιπόν ακριβώς αυτό το νήμα το ερυθρό που συνδέει το πρώτο κεφάλαιο με το τελευταίο. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα των εθνικών διδακτικών προγραμμάτων ιστορίας. Προσπαθούμε εμείς να εμπλουτίσουμε αυτή τις διαδικασίες τις εκπαιδευτικές δεν μπορούμε να είμαστε φιλόδοξοι βέβαια υπερβολικά αλλά κάνουμε προτάσεις ήδη ε, για τους ε, καθηγητές ε, με 150 καθηγητές μέσω του προγράμματος Euroclio. Είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν και η πλειοψηφία των καθηγητών είπαν ότι αυτή η διαδικασία ήταν μια θετική διαδικασία και μια επιπλέον ένα εκπαιδευτικό στοιχείο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν και στα εθνικά τους προγράμματα. Συγγνώμη, κάτι άφησα. 350.000 ε, ε, ε, το χρόνο γιατί είναι μικρό το κτίριο βέβαια για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να έρχονται στις Βρυξέλλες μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορες προσφορές και μία ώρα και 20 λεπτά αρκεί για να περάσει κανείς από την έκθεση και να κρατήσει τα βασικά μηνύματα. Αν κάποιος θέλει να μείνει περισσότερο μπορεί να μείνει τρεις μέρες, μια εβδομάδα μα θέλει και να έρχεται όσο συχνά θέλει. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ λοιπόν και την ε, Διευθύντρια του οίκου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Πρόκειται για κάτι λοιπόν το οποίο ανήκει σε όλους, πρόκειται για κάτι το οποίο είναι ανοιχτό, δεκτικό και εξελίσσεται συνεχώς και θα πρέπει οι διαδικασίες αυτές της ανοικοδόμησης του συνόλου της ιστοριογραφίας πρέπει να παραμείνει σε συνεχή αλλαγή, δεν είναι ένα τελειωμένο προϊόν, αλλά είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει να διατηρήσουμε την ιστορία και τις καταβολές που όλοι θέλουμε. Εύχομαι λοιπόν να σας δω ε, το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την παρουσία τους. Τελειώσαμε το θέμα αυτό. Πριν από το τέλος έχουμε ένα ακόμη θέμα παρακαλώ 5 με 10 λεπτά. Eh, Πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, σε πέντε λεπτά να προσπαθήσουμε να τελειώσουμε, αλλά να μην φύγει όλος ο κόσμος. Ε, το θέμα αυτό ε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό σημαντικό θα είναι πριν από, την από τα επίσημα εγγένειες 17 Νοεμβρίου να κάνουμε μια επίσκεψη. Λοιπόν, το τελευταίο σημείο αφορά την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Είναι σημαντικό το σημείο αυτό πιστεύω εγώ είμαι συντάκτρια και κυρίως όσον αφορά την έμφαση στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής CPRD του ΟΗΕ. Είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό, διότι θέλω να υπενθυμίσω συναδέλφους ότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη συνθήκη των Ευρωπαϊκών ε, των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία τέθηκε σε ισχύ 22 Ιανουαρίου του 2011 και είμαστε η πρώτη περιφερειακή οργάνωση που επικύρωσε συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Ηνωμένα Έθνη εφαρμοστεί από το 2014 και να σας υπενθυμίσω ότι μετά από αυτό ε, τα Ηνωμένα Έθνη τον Απρίλιο του 2015 παρουσίασαν μια λίστα εκκρεμών προβλημάτων τα οποία θέλουν διευκρινήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε ένα έγγραφο με απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, για αυτό το λόγο το Μαΐο του 2015 ε, υιοθετήσαμε εμείς εδώ ένα ψήφισμα για τη λίστα αυτή προβλημάτων τέλος σήμερα εδώ θα μιλήσουμε για τις καταληκτικές παρατηρήσεις του Σεπτεμβρίου 2015 της Επιτροπής CPRD του ΟΗΕ. Οπότε αυτό το σχέδιο αφορά τα συμπεράσματα της Επιτροπής του ΟΗΕ μετά από τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα έχετε δει το σχέδιο εκθεσής μου. Ε, οι παρατηρήσεις μου αναφέρονται κυρίως στο ζήτημα της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά όχι μόνο αλλά και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό τρεις διαφορετικές πτυχές ε, της πολιτικής ένταξης να υπενθυμίσω ότι πρόκειται περί δικαιωμάτων και όχι επιλογών να δεσπίζονται από τα άρθρα της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών 19, 24 και 30 και κυρίως όσον αφορά την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης λόγω αναπηρίας, αναπηρίας και εδώ ζητάμε από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τα μέτρα που διασφαλίζουν την ίση πρόσβαση στον πολιτισμό και στον αθλητισμό και στην εκπαίδευση να επισημάνω ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο αίτημα από κάποιους συνομιλητές να το ζητήσουμε στεναρά και στα ευρωπαϊκά σχολεία, στο καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων, όπου δεν διασφαλίζεται πάντα η πρόσβαση των ε, ατόμων με αναπηρία. Δεύτερον, καλύτερη χρήση των ε, Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών ε, Ταμείων και των Ευρωπαϊκών Επενδυτικών Ταμείων για την υποστήριξη των υποδομών πρόσβασης ε, των ατόμων με αναπηρία αλλά για να είναι και πιο προσπελάσιμα τα δικά μας προγράμματα, το Creative Europe, το Erasmus κτλ. Τίθε επίσης το ζήτημα της ένταξης των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα σχολικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα από παιδιά έως ενήλικες, είτε αναφερόμαστε σε σωματικές είτε σε πνευματικές αναπηρίες. Το τρίτο που αναφέρουμε είναι επαρκή κατάρτιση των διδασκόντων. Συχνά παρατηρούμε αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία από αυτές τις υπηρεσίες, δεν έχουν επαρκή πρόσβαση. Θα πρέπει λοιπόν να δράσουμε ώστε οι διδάσκοντες ε, ε, να μπορούν να υποστηρίξουν άπαντες στις τάξεις ε, έχοντας προετοιμαστεί και καταρτιστεί επαρκώς. Το άλλο σημείο αφορά την κινητικότητα ε, τα άτομα με αναπηρία όπως γνωρίζετε πολύ περισσότερο στο παρελθόν ε, ε, προσχωρούν στα προγράμματα κινητικότητας των φοιτητών. Το άλλο πρόβλημα είναι η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων για τα άτομα με αναπηρία και έτσι λοιπόν αυτό που είναι σημαντικό για μας ε, με την έγκριση της συνθήκης του Μαρακές που θέλει να διευκολύνει την πρόσβαση σε διάφορα έργα για άτομα με προβλήματα όρασης και σε όλα τα ψηφιακά μέσα γενικότερα και στις διάφορες ιστο, ιστοσελίδες ε, η προσφυγή στις assisted technologies όπως ονομάζονται ώστε να δο, ε, διευρυνθούν οι ευκαιρίες αλλά και η μάχη που πρέπει να γίνει με πολλά κριτήρια και κανόνες ώστε να καταπολεμήσουμε το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και την παρενόχληση στον κυβερνοχώρο. Έχουμε και πολλές περιπτώσεις αυτοκτονίας ε, στον κυβερνοχώρο λόγω τέτοιων περιστατικών. Ε, πρόκειται για ένα δραματικό φαινόμενο. Και τέλος, έχουμε ζητήσει από την Κομισιόν να ξεκινήσει μια εξτρατεία ευαισθητοποίησης Ε, δυνάμει του χάρτη, της ε, συνθήκης, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την ευαισθητοποίηση περί της ε, αναγκαιότητας προφύλαξης αυτού του δικαιώματος. καθώς και για να επισημάνουμε την αναγκαιότητα να γνωρίζουν τα άτομα με αναπηρία όλα τους τα δικαιώματα στην Ευρώπη. Αυτά τα σημεία έχω επισημάνει εγώ. Φυσικά είμαι διατεθειμένη να υποβάλω συμβαστικές τροπολογίες ε, αλλά είμαι βέβαιη ότι θα υποβάλλετε και εσείς να υπενθυμίσω προθεσμία για, αυτές, για τις τροπολογίες σας είναι 5η-25 Φεβρουαρίου στις 12 ψηφοφορία στην Επιτροπή 19 Απριλίου στην επί αρμόδια επιτροπή που είναι η ΕΜΠΛ ψηφοφορία στις 30 Μαΐου του 2016 αν δεν υπάρχουν προβλήματα έχουμε 5 λεπτά νομίζω ε. Ε, έχουν ζητήσει οι σκιώδεις ε, το λόγο και συνάδελφος Κομοντίνη α συγγνώμη αλλάξατε θέση Κομοντίνη Νταμπρόφσκι Εύανς Φεράιν. Ωραία ευχαριστώ Ευχαριστώ ένα από τα βασικά σημεία τα οποία θα ήθελα να θέσω είναι αφού σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση της πρότασής σας τα σημεία τα οποία ήδη παρουσιάσατε έχουν μεγάλο βάρος. Πιστεύω ότι υπάρχει εδώ μια αρχή η οποία είναι θεμέλιο ή μάλλον δύο αρχές που θα έλεγα είναι θεμέλια της πρότασής μας. Πρώτον θα πρέπει να βελτιώσουμε το πνεύμα της σύμβασης. Βασικός στόχος της συγκεκριμένη σύμβασης είναι να προκαλέσουμε μια πολιτιστική αλλαγή στον τρόπο που βλέπουμε την αναπηρία, ε, όχι ειδικά για το πρόσωπο αλλά το εμπόδιο ε, της αναπηρίας ε, να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε λόγω όταν προκαλείται από το περιβάλλον. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στη γνωμοδότησή μας το δεύτερο, η δεύτερη θεμελιώδης αρχή την οποία πρέπει να συμπεριλάβουμε και νομίζω ότι έχετε κάνει τη σωστή αρχή είναι να προσπαθήσουμε έτσι ώστε όλες οι αρμοδιότητες αυτής της Επιτροπής να υπογραμμιστούν στην έκθεση. Εκτιμώ ήδη τα σχόλια τα οποία κάνατε για την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και την παιδεία και τον πολιτισμό λοιπόν ε, νομίζω ότι μπορούμε να τα υπογραμμίσουμε ακόμα περισσότερο στο εσωτερικό της γνωμοδότησης και δεν θα πρέπει να εξαιρέσουμε θα έλεγα αναφορές για τους νέους, τα πολιτικά μέτρα για τους νέους και τα μέσα ενημέρωσης. Ε, στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών υπάρχουν στοιχεία τα οποία άπτονται άμεσα των δικών μας αρμοδιοτήτων πρέπει να ανταορίσουμε καλύτερα και να αντιδράσουμε σε αυτά και υπάρχουν και κάποιες άλλες παρατηρήσεις έμεσα αναφερόμενες στις δικές μας αρμοδιότητες και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε σε βάθος. Ε, ένα από τα θέματα αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν και μας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προχωρήσει στο λεγόμενο mainstreaming των θεμάτων αναπηρίας και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να χαρακτηρίζει το σύνολο των αρμοδιοτήτων μας. Υπάρχουν φυσικά πάρα πολλά τα οποία μένει να γίνουν ιδιαίτερα σε σχέση με τη χρήση της εκπαίδευσης του αθλητισμού και του πολιτισμού γιατί έχουμε και την πλευρά της ε, προσπάθειας να καταστήσουμε τους τομείς αυτούς προσβάσιμους στους ανθρώπους με αναπηρίες αλλά έχουμε και τομείς οι οποίοι μπορεί από μόνοι τους να συνεισφέρουν στο να ξεπεραστούν τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν σε επίπεδο πολιτιστικό, σε επίπεδο αντίληψης. Να υπογραμμίσουμε τις δυσκολίες πρόσβασης των ανθρώπων με αναπηρία και να κάνουμε και προτάσεις έτσι ώστε να αντιστρέψουμε τα αρνητικά αυτά χαρακτηριστικά και να καταστήσουμε εφικτές τις λύσεις. Ένα πάρα πολύ καλό σχόλιο θα έλεγα, πρόταση την οποία ήδη έχετε κάνει είναι του ότι οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές να είναι σωστά εκπαιδευμένοι για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους θεμάτων. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που ήθελα να θέσω σήμερα. Ε, θα ήθελα επίσης να συνεχίσουμε την συνεργασία μαζί σας κυρία Κώστα και με τους άλλους σκιώδεις. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή γνωμοδότηση για τους ανθρώπους με αναπηρίες. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και για τις προτάσεις ο κύριος Τσαμπάσκι. Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Τσαμπάσκι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την Πρόεδρο για την παρουσίαση της νομοδότησης αυτής για τους ανθρώπους με αναπηρίες είναι σωστή ιδέα για την έκθεση αυτή, μια έκθεση ιδέας πρωτοβουλίας. Η Χέλγκα Στίβενς ξέρετε ότι είναι ιδιαίτερος φιλόδοξη στον τομέα αυτό και δραστήρια. Υπάρχουν πολλοί τομείς τους οποίους πρέπει να καλύψουμε όπως η αναθεώρηση της υπάρχουσας διαδικασίας ε, στο εσωτερικό των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα των διακρίσεων εις βάρος των ανθρώπων με αναπηρίες ε, πρέπει να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα στον τομέα των παιδιών και των γυναικών με αναπηρίες αλλά και στους υπόλοιπους τομείς. Είναι δύο οι αρμόδιες επιτροπές και ακόμα και κάποιες άλλες επιτροπές ε, θα πρέπει να γνωμοδοτήσουν. Θα είναι μεγάλη σε μέγεθος η έκθεση αλλά θα πρέπει να παραμείνει σωστά στοχευμένη. Αυτά τα οποία προτείνει η κυρία Κώστα είναι οι σωστές κατευθυντήριες γραμμές και ελπίζω να υιοθετηθεί το ταχύτερο δυνατόν να επικυρωθεί μάλλον η υιοθέτηση της συμβάσεως του Μαρακές ή της συνθήκης καλύτερα του Μαρακές και θα πρέπει επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό μόντζουλ για την σωστή κατάρτιση των εργαζομένων που θα βοηθήσει την ένταξη των ανθρώπων με αναπηρίες και, την, ε, ε, και τα επιμέρους δικαιώματα όπως την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την ε, βοήθεια για την υπέρβαση εμποδίων κτλ. Evans, ευχαριστώ. Να πω ότι η έκθεση αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και ότι υπάρχουν πολλές κοινοβουλευτικές επιτροπές που θα γνωμοδοτήσουν δείχνει το μέγεθος και τη σημασία της. Πρέπει να υπογραμμίσουμε τα θέματα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, ε, του αθλητισμού. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Για την κοινωνική πτυχή ξέρω ότι το ζήτημα Rails ε, που συνεργάζεται με ΜΚΟ έχει αθετήσει αυτό το κοινωνικό μοντέλο εξετάζοντας όχι μόνο τις αναπηρίες αλλά και το πώς ε, τα εμπόδια μπορούν να υπερπηδηθούν, τα εμπόδια για την ισότητα. Ο πολιτισμός φυσικά μπορεί να βοηθήσει να υπερπηδήσουμε αυτά τα εμπόδια ε, μέσω πολιτιστικών αλλαγών. Κάτι που ήθελα να επισημάνω ιδιαίτερα σχετίζεται με το διαδίκτυο, τις διαδικτυακές υπηρεσίες κτλ. Στη δική μου εκλογική περιφέρεια το 38% των ατόμων με αναπηρία δεν μπορούν να συνδεθούν online. Ένα πράγμα λοιπόν που λέμε ε, ότι θέλουμε να κάνουμε στην Ουαλία είναι να απασχολήσουμε εθελοντές που θα εκπαιδεύσουν όλο και περισσότερους ανθρώπους ε, για να αποκτήσουν συνδεσιμότητα και προσβασιμότητα. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που αναφέρατε. Ε, επίσης ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτή την εκστρατεία ευαισθητοποίησης. Επίσης και το ζήτημα των γλωσσών μειονοτήτων είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη Περιμένουμε υπομονησία λοιπόν να συνεργαστούμε για όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τις προτάσεις σας. Παρακαλώ, Σαμπίν Φερχαΐν. Πολλά λέχθηκαν ήδη. Γι' αυτό θα έρθω στην παράγραφο 4 του σχεδίου. Επιθυμώ να τονίσω ότι αυτό που ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει ήδη κάνει. Άρα πρέπει να προσέχουμε λιγάκι τα αιτήματά μας να μην έρχονται καθυστερημένα. Ήδη υπάρχουν οι διαπραγματεύσεις στον τριμήρη διάλογο για το θέμα Sensibility in Public Sector Websites όπου εξηγούμε ποια κριτήρια πρέπει να θεσπιστούν ώστε να είναι προσβάσιμες τέτοιες ιστοσελίδες και οι αναπήρους. Το ίδιο ισχύει και για το Accessibility Act που είχε ήδη υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως σχέδιο νομοθετήματος πέρσι. Και αν θα μπει πλέον στην κοινοβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να δούμε αν θα χρειαστεί να κάνουμε γνωμοδοτήσεις ως Επιτροπή Πολιτισμού. Διότι στην συζήτηση για την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων του δημόσιου τομέα έχουμε ήδη ε, έχουν ήδη γίνει τα σχετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συναδέλφοι. Πολλές συμβουλές δώσατε. Πολύ χρήσιμα σχόλια. Ίσως η Κομισιόν να θέλει το λόγο. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Παρακαλώ. Και μετά θα κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήθελα παρά να πω ότι η Κομισιόν καλωσορίζει όλα τα σχόλια και το σχέδιο κειμένου που παρουσιάσατε. Συμφωνούμε φυσικά τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει οπωσδήποτε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς και ειδικότερα αυτών που έχουν ειδικέ ανάγκες. Από άποψη εκπαίδευση συνεργαζόμαστε με συναδέλφους εντός της Κομισιόν ε, ώστε να υπάρξει κάποια καλή συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών για να συμβάλλουμε στους διάφορους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία μέχρι το 2020 και εκεί υπάρχει ένα θέμα που προωθεί την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και τη διαβίου μάθηση για άτομα με αναπηρία. Είναι λοιπόν συνεχές το έργο μας. Θα παρατηρήσατε επίσης όταν συζητούσαμε για την κοινή για το σχέδιο κοινή έκθεση νωρίτερα ότι ένα από του τομεί προτεραιότητα και ένα από τα συγκεκριμένα ζητήματα που θέλουμε να μελετήσουμε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και άλλου ενδιαφερομένου είναι το να διασφαλίσουμε ότι έχουμε ε, ε εκπαίδευση υψηλή ποιότητα χωρίς αποκλεισμούς ε, με τη συμμετοχή όλων και των ατομών με αναπηρία. Αποτελεί λοιπόν κομμάτι όλων των επέδων εργασία μα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίση, ε, συνεργαζόμαστε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Άτομα με Ανάγκε και την εκπαίδευση χωρί αποκλεισμού, με τακτικέ αναθεωρήσει και παρακολούθηση των εξελίξεων στα κράτη-μέλη. Προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε διαρκώ ε, συντονισμένοι και να αλληλοϊποστηριζόμαστε όσον αφορά την κατανόηση των εξελίξεων και των προκλήσεων που απομένουν στα διάφορα κράτη-μέλη με τον οργανισμό αυτό για τα άτομα με ειδικέ ανάγκε. Και όπω αναφέρετε, ορισμένοι από εσά, τέλο το Erasmus Plus. Και εκεί προσπαθούμε να κάνουμε μια διαρκή προσπάθεια βελτίωσης της προσβασιμότητας ε, για φοιτητέ ε, με αναπηρία, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις ε, για τη συμμετοχή όσον αφορά την οικονομική στήριξη ουσιαστικά των ε, ατόμων με αναπηρία. Αλλά πέραν της, ε, του σκέλους της κινητικότητας στο πρόγραμμα υποστηρίζουμε και διάφορα άλλα προγράμματα με διάφορους ενδιαφερομένους ώστε να εντοπίσουμε κάποιες καλές πρακτικές μέσω της ανταλλαγής απόψεων για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και την Κομισιόν για τις συστάσεις και προτάσεις, τις πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις. Ε, τα όσα είπε η κυρία Κομοντινή και οι υπόλοιποι. Πρέπει να υπογραμμίσουμε φυσικά τη βασική αρχή, όπως είπε και η κυρία Evans, ότι πρέπει να βρούμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία αντί να αντιμετωπίζουμε τα άτομα αυτά ως ε, άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, να άρουμε απλά τα εμπόδια που τους εμποδίζουν. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, κάτι πολύ σωστό θεωρώ, ε, καταθέτω και τροπολογίες εγώ γι' αυτό, όλοι οι χώροι, σε όλους τους χώρους για τους οποίους έχουμε αρμοδιότητα, υπάρχουν άλλες δύο πτυχές. Ε, ο εθελοντισμός ενεργός, όχι μόνο παθητικός, αλλά και η πολιτιστική, δημιουργική και καλλιτεχνική εκπαίδευση στην Ευρώπη. Σκέφτομαι με το θέατρο, με συμμετοχή ατόμων με αναπηρία. Ε, και έτσι δημιουργούνται και δίκτυα. Συμφωνώ με τα ζήτημα αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας ε, για τα σημεία όπου δεν καλύπτει τα θέματα που μας απασχολούν εμάς Υπάρχει και κάποιες ιδιαιτερότητες, μιλήσαμε για το Μαρακές, ε, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και το ζήτημα της ε, ε, Οπότε να υπάρξει μια διεθνής αναγνώριση όλης αυτής της προσέγγισης και για την νοηματική Επίση, θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε και στα διάφορα προγράμματα όπω το Εράσμου ε, να εφαρμόζονται όλα αυτά που προβλέπονται. Συμφωνώ φυσικά όσον αφορά τι διάφορε ηλικίε και τα φύλλα, τι διάφορε ευαισθησίε και τι διάφορε πτυχέ, ε, και σημειώνω τα όσα είπε και η συνάδελφο κυρία Φερέιεν για τι πτυχέ που έχουν ήδη επιληθεί στον τριμερή διάλογο αλλά για παράδειγμα το θέμα τη πρόσβαση, στη δυνατότητα χρήση του διαδικτύου όχι μόνο η πρόσβαση λοιπόν στο διαδίκτυο, αλλά και η πρακτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ιταγένειας από αυτά τα άτομα είναι σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να τα μελετήσουμε όλα αυτά σε συνεργασία μεταξύ μας. Εδώ κλείνει αυτό το εντατικό προϊόν, πρωινό εργασίας. Ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Θα συνεχίσουμε στις 3 ακριβώς. Και σήμερα έχουμε μια γεμάτη μέρα με το παρατηρητήριο σε σχέση με την παραβίαση των, ε, διανοητικών δικαιωμα... δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τις διάφορες εκθέσεις για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους. Καλή σας όρεξη. Τα λέμε στις 3.